Item number five. We now proceed... Συνάδελφοι, πέντε, να περάσουμε στην πρώτη εξέταση της ε, σχεδίου σύστασης ε, για τα θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια σχετικά με την προάσπιση τη ακαδημαϊκή ελευθερία στην εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριο Καν είναι ο εισηγητή μα, ο οποίο μόλι και κατέφτασε. Watch. Αν ε, είσαι έτοιμο, πάρε το λόγο. Thank you, Chair, and thank you for your... Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιπλέον υπομονή που δείξατε εκ μέρους της ομάδας Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση για την υπεράσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ότι ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντρικού λάνκασιερ πριν γίνω Ευρωβουλευτής και είναι πολύ ανήσυχοι οι συνάδελφοί μου για τις συχνές επιθέσεις που δέχεται η ακαδημαϊκή κοινότητα σε όλη την Φίλιο. Ε, φυλακίζονται, λογοκρίνονται, ε, ακόμα και δολοφονούνται ε, επειδή ακριβώς διδάσκουν και δηλώνουν. Σε πάρα πολλά κράτη υπόκεινται σε λογοκρισία γιατί υπάρχουν πολιτεύματα τα οποία προσπαθούν να καταπιέσουν την ελευθερία του λόγου και δεν καταστρέφει μόνο ζωές, αλλά δεν επιτρέπει και σε όσους το χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στη γνώση των εμπειρογνωμόνων. Δεν γίνεται δημόσια συζήτηση και όλα αυτά περιορίζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και παρακολύουν την κοινωνική ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα πήγα ως ε, μέλος ε, αντιπροσωπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα πως γίνεται μια επίθεση στην ελευθερία του λόγου με μια χωρίς προηγούμενο ε, δίωξη ακαδημαϊκών. Και βέβαια μαθαίνουμε κάτι αντίστοιχο για την Κίνα. Στοχευμένες επιθέσεις στο Ιράν, Νικαράγουα, πιέσεις που όλα αυξάνονται στις ΗΠΑ και επίσης απειλές κατά των ακαδημαϊκών Ινστιτούτων και στη Ρωσία αλλά και στην Ουγγαρία που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η UNESCO μιλά για μια ελευθερία θεμελιώδη χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς ε, καμία ε, επιταγή και με την ελευθερία και έρευνας και διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και ελευθερία έκφραση λόγου οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε σύστημα να ε, εργάζεται κανείς. Ελευθερία από την θεσμική λογοκροσία και ελευθερία συμμετοχής σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δυστυχώς πάντως όλα αυτές, όλες αυτές οι παραβιάσεις αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος πολύ σπάνια αναφέρονται στα πλαίσια των παραβιάσεων των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων και δεν τυχάνουν της ίδιας αναγνώρισης με τα υπόλοιπα. Έχουμε μια πολύ συχνή παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων τα οποία επαναλαμβάνω ε, δεν ε, συζητιώνται. Είναι ένα ε, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή μας και να λύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα που είναι η αναγνώριση και η συζήτηση αυτών των προβλημάτων. Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία κάνουν πολύ καλή δουλειά και όπου παρακολουθούν παραβιάσεις και διώκουν όσους... ασκούν αυτές τις ποιότητες, Αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει πιο διαδεδομένο και να έχουν και οι ίδιοι οι φοιτητέ τη δικαίωμα καταγγείλες. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε η ηγετική θάση σε αυτή τη ε, δράση και να προωθήσουμε εμείς την ακαδημαϊκή ελευθερία παγκόσμια. Στην έκθεση αυτή που είναι πρωτοβουλία δίνουμε κάποια συστάσεις για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα τροτά άτομα και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα αναφοράς, περισσότερη ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση, διάλογο και την κατανόηση που θα αποφύγει τέτοιου είδους απειλές σε όλη την φίλη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ που με ακούσατε συνάδελφοι και με μεγάλη χαρά ε, συνεδριάζουμε με τους ε, συναδέλφους, τον κύριο Τάνοκ, τον κύριο Τσούκ, την Άντρια και τον κύριο Μπρούκνερ για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ επαναλαμβάνω που μου δώσατε το χρόνο και το γεγονός πως με περιμένατε γιατί στο πρωί καθυστέρησα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας. Προχωρούμε σε σύντομη συζήτηση. Έχω πέντε συναδέλφους εγγεγραμμένους. Σιουκ, Καστάλτο Επιτιδέος. Μήπως ε, ξέχασα κανένα όνομα. Όχι. Ωραία. Δύο λεπτά παρακαλώ ο κάθε ένας και αρχίζουμε με την κυρία Μποσκόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα αλλάξω γλώσσα τώρα από τα αγγλικά. Θα μιλήσω ουγγρικά και σας παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Είναι, η ανθρώπινη περιέργεια είναι ένα προσόν, είναι αυτό που μας ε, επιτρέπει και την πρόοδο. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ελευθερία της ε, πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής ε, παιδείας είναι σε μεγάλο κίνδυνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Για αυτό το λόγο σε πολλές χώρες δηλαδή. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Ορισμένα πράγματα γίνονται αποδεκτά, αλλά δεν γίνονται σε άλλες χώρες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι ωστόσο σημαντικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς ωστόσο να πολιτικοποιήσουμε υπερβολικά το θέμα, διότι αυτό μπορεί να έχει και αντίθετα αποτελέσματα. Ο συνάδελφός μου προηγουμένως μίλησε για προβλήματα χωρών του τρίτου κόσμου και εκεί έβαλε μαζί και την Ουγγαρία. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ούτε θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα μου στην ε, έκθεση αυτή. Μιλήσατε για το Κέντρο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με την ακαδημαϊκή ελευθερία. Όταν μιλούμε για ακαδημαϊκή ελευθερία δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ποιότητα εκπαιδεύσεως στην Ευρώπη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της παιδείας. Η ενσωμάτωση φοιτητών που δεν διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και η ενσωμάτωση διδασκόντων από ξένες, ε, παραδοσιακές, από ξένες μάλλον πολιτιστικές παραδόσεις επίσης δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Από την άλλη μεριά έχουμε και αυτή τη φυγή εγκεφάλων που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω όμως και τον συναδελφό μου, σε ποιες στατιστικές βασίζετε τις δηλώσεις σας που περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Κιουτσούκ. Θα είμαι σύντομο κύριε Πρόεδρε. Πρώτα συγχαίρω τον αγαπητό μου συνάδελφο Ουαζίτ Καν για τη σημαντική εργασία που έχει ε, βάλει στην ε, ισορροπημένη αυτή έκθεση για την προάσπιση τη ακαδημαϊκή ελευθερία, τη εξωτερική δράση τη Ένωση. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι από τα πιο σημαντικά δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω κάνει και εγώ, ε, είμαι και εγώ σκιώδη και είναι σημαντικό, ξαναλέω, για τις εξωτερικές δράσεις. Πρέπει να ενταθούν οι διπλωματικές οι ε, προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή ελευθερία με αποφυγή και αποτροπή επιθέσεων κατά των ακαδημαϊκών θεσμών. Γιατί κινδυνεύουν και οι φοιτητές οι ίδιοι και οι καθηγητές. Εγώ θα καταθέσω και ορισμένε τροπολογίες στο κείμενο. Γενικά όμως πιστεύω ότι η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη αποτροπής επιθέσεων κατά του καδημαϊκού επίπεδου. Σας ευχαριστώ. Φάμπιο Καστάλντο της ομάδας EFDD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για την soft power, για την ήπια δύναμη που είναι ένας από τους μοχλούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της, κυρίως στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την έκθεση που συντάσσει ο φίλος μας ε, Ουαζίτ Καν. Είναι πολύ σημαντικό η ελευθερία των πανεπιστημιακών να είναι εγγυημένη, να έχουν ένα χώρο ελευθερίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Βλέπουμε ωστόσο ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ο πανεπιστημιακός κόσμος βρίσκονται υπό μεγαλύτερη απειλή διαρκώς και περιορισμούς από εξωτερικούς παράγοντες. Υπάρχουν πα, πάμπολοι πανεπιστημιακοί στις φυλακές, μόνο και μόνο επειδή εξέφρασαν την άποψή τους. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει προσπάθεια να προτραπούν οι, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να επιτρέπουν την ελευθερία έκφρασης. Θυμίζω το παράδειγμα της Κίνας, όπου πολλές χιλιάδες πανεπιστημιακοί βρίσκονται στις φυλακές λόγω των απόψεών τους. Και μιλώ πάντοτε για πανεπιστημιακούς δασκάλου και φοιτητέ. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε, αυτή, σε αυτόν τον περιορισμό και πρέπει να, ε, να βοηθήσουμε να τους καταπολεμήσουμε. Ο ρόλος επίσης που μπορούν να παίξουν οι αρχές, ακόμα και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτόν πρέπει να τον εξετάσουμε, διότι η πίεση ασκείται σε όλα τα επίπεδα η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της εκφράσεως αποτελούν τα θεμέλια αυτών των ελευθεριών που όλοι έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε και είναι και οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν και τις εξωτερικές μας σχέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις θεμελιώδεις αυτές ελευθερίες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελευθερία της σκέψεως, Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Θα ήθελα να προχωρήσουμε σε περισσότερο βάθος. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και πίεση χρόνου. Πάντως ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ τον κύριο Καστάλδο, ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία, επειδή ακριβώς είναι συνειφασμένη με την ελευθερία της σκέψης και της εκφράσεως, είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να διδάξουμε τους νέους επιστήμονες να έχουν δημοκρατική αντίληψη και δραστηριότητα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η προσπάθεια που καταβάλει ο εισηγητής και γι' αυτό ακριβώς το συγχαίρω. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να προσέξουμε πριν καταδικάσουμε την οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των ελευθεριών στις τρίτες χώρες την δική μας παραβίαση, και όταν λέω δική μας εννοώ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παραβίαση αυτής της ελευθερίας στα πανεπιστήμια. Αναφέρομαι σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πρόσφατα σε κάποιο πανεπιστήμιο της Σουηδίας. Κάποιος καθηγητής είπε το αυτονόητο, ότι οι γυναίκες και οι άντρες γενεολογικά έχουν διαφορές. Ο άνθρωπος αυτός έγινε αντικείμενο διώξεων, του ζητήθηκε να αναιρέσει και κινδυνεύει να απολυθεί από τη θέση του. Αυτό δεν προάγει την ελευθερία. Πριν λοιπόν καθαρίσουμε την αυλή του γείτονα, ας αποφασίσουμε να καθαρίσουμε πρώτα την αυλή τη δική μας. Ευχαριστώ. Thank um, Είναι προφανές είναι προφανή μάλλον η σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερία. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, τον Μεσαίωνα η Σορβόνη είχε ειδικό καθεστώ έξω εδαφικότητα. Κάντε συγκεκριμένες προτάσεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ώστε η έκθεση να μην είναι απλό ευχολόγιο, αλλά να ε, διασφαλίζει πραγματικά την ελευθερία αυτή. Και η μεγαλύτερη ελευθερία θα ήταν να έχουν τα πανεπιστήμια ένα είδος καθεστώτος όπως έχουν τα, οι πρεσβείες. Κάνω την πρόταση αυτή και ελπίζω ότι θα τη δεχτείτε και ότι πράγματι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να προοδεύσει η ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή ελευθερία. Όταν τώρα ένα πίσω από το πανεπιστήμιο διακόπτει ο κύριος Μακαλίστερ, διακόπτει φαίνεται πως υπάρχει ένα πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση. Μπορείτε να το κοιτάξετε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά δεν λειτουργεί η μετάφραση. Κανείς δεν μεταφράζει μεταξύ γαλλικών και αγγλικών, ρωτάει ο κ. Σαφχάουζε. Α, ωραία, φαίνεται πως διορθώθηκε. Ξαναρχίζω, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη πρόταση λοιπόν που κάνω στο συναδελφό μου είναι να εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις και μια συγκεκριμένη πρόταση είναι να χορηγηθεί στα πανεπιστήμια το ίδιο καθεστώς όπως για παράδειγμα ε, οι πρεσβείες. Και ξαναλέω ότι στο, μεσ, στο μεσαίωνα ε, το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης ε, έχερε του καθεστώτος της εξοδαφικότητας και ένα είδος ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας τόπος ιερός. Είχε ένα άβατο. Ε, αυτά για την ελευθερία. Τώρα, όταν το πανεπιστήμιο όμως, για τον κύριο Σόρος, γίνεται τόπος πολέμου και οργάνωσης και οργάνωσης αγώνα κατά ενός νόμιμου κράτους, ε, δεν είναι το ίδιο πράγμα, το πανεπιστήμιο και ο κύριο Σόρος είναι αυτός που μετασχηματίζει, μεταμορφώνει το πανεπιστήμιο σε όργανο αγώνα κατά ενός νόμιμου καθεστώτος. Δεν πρέπει λοιπόν να καταδικάζουμε τον κύριο Ορμπάν, αλλά τον κύριο Σόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο ως όργανο πολιτικής προπαγάνδας. Πρόκειται για έσχος. Και θα προσθέσω μάλιστα ότι θα είναι σωστό να μελετηθούν τα, οι σχέσεις του κύριου Σόρος με εξωτερικές δυνάμεις και καμιά φορά και με το οργανωμένο έγκλημα. Υπό τις συνθήκες αυτές νομίζω ότι πρέπει αφενός να ενισχυθεί το καθεστώς των πανεπιστημίων και της πανεπιστημιακής ελευθερίας, αλλά όχι να, χώνεται μέσα σε όλα αυτά και την Ουγγαρία. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σαφχάουζε. Μάλιστα. Η κυρία Αλιό Μαρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως παλαιά πανεπιστημιακή θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Καν και να τον συγχαρώ, να πω ότι στηρίζω το σύνολο της εκθέσεως, θα επισημάνω κάτι και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι και νομίζω και εσείς, εσείς ο ίδιος κύριε Καν ε, το θίξατε και μιλώ για την σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή ελευθερία και στην ελευθερία εκφράσεως. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη ελευθερία εκφράσεως, διότι βλέπουμε σε ορισμένες από τις χώρες μας το πρόβλημα της εκφράσεως μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο, απολογία ε, της τρομοκρατίας, απολογία του σεξισμού, άρνηση ε, ιστορικών γεγονότων όπως το ολοκαύτωμα και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη. Η πανεπιστημιακή ελευθερία είναι και η ελευθερία να εκφράζεται κανείς. Ναι, αλλά πρέπει να κάνει μια επιλογή. Μέχρι πού φτάνει η πανεπιστημιακή ελευθερία. Οι θέσει των χωρών μας είναι διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό κρίνω ότι μια συζήτηση είναι αναγκαία. Η συζήτηση αυτή είναι αναγκαία διότι θα εξυπηρετήσει και στην ενίσχυση του περιεχομένου της εκθέσεώς σας. Ε, ό,τι ξαναλέω πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Άλλος κανείς, σας παρακαλώ, που θα ήθελε να ομιλήσει. Δεν βλέπω, δεν βλέπω το όνομά σας. Ορίστε. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς την κυρία Αλιό Μαρή. Ποιο θα αποφασίσει τι επιτρέπεται να λέγεται μέσα στα πανεπιστήμια και ποιο όχι. Και, και συγγνώμη, και τι όχι. Ε, η, η, η Μισελ Αλιομαρή είπα ότι θα πρέπει να διεξαχθεί μια συζήτηση, πιθανότατα μάλιστα εδώ, η πανεπιστημιακή ελευθερία επιτρέπει να λέγεται οτιδήποτε ή υπάρχουν κάποια όρια. Αυτό εξαρτάται από την κάθε χώρα. Δεν νομίζω ότι οι θέσεις μπορούν να είναι οι ίδιες. Αυτό που λέω είναι ότι στην έκθεση δεν μπορεί να βγει εκτός παρενθέσεως, ας πούμε, η, ε, υπόθεση αυτή. Αλλά πρέπει να περιληφθεί. Μακάλιστερ αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να βρουν το λόγο. Είχαμε προβλέψει 15 λεπτά για την συζήτηση αυτή και θα ήθελα να κρατήσουμε το χρονικό αυτό όριο, διότι έχουμε και άλλα θέματα. Θα διεξαχθεί ούτω ή άλλω και άλλη συζήτηση όπου μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει. Θέμα υπαριθμών 6 έχουμε ήδη 15 λεπτά καθυστέρηση. Έρχομαι λοιπόν στην έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Σερβία και μετά για το Πέδιο. Για τη Σερβία είμαι ο ίδιος εισηγητής, θα σας ενημερώσω λοιπόν σύντομα. Η πρώτη εξέταση έγινε στις 21 Έκτου, η προθεσμία κατά καταθέσεως τροπολογιών ήταν 24 Αυγούστου. Εν τέλει συνελέχθησαν 239 τροπολογίες, 86 λιγότερες από το 2016 και αν θυμάστε καλά το 2017 δεν έγιναν τα σχετικέ εκθέσεις. Οι περισσότερες ε, τροπολογίες αναφέρονται σε δικαιώματα των μειονοτήτων, σε συνεργασία, ελευθερία του τύπου κλπ. Την τρίτη το απόγευμα διεξήχθη μια καρποφόρα συνάντηση με τους γιώδεις συγητές, όπου όλοι συμφώνησαν το ψήφισμα να γίνει όσο γίνεται πιο ισορροπημένο, κάτι το οποίο νομίζω επιτύχαμε είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η Σερβία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να υπάρξει και χώρος για να αντιμετωπιστούν κάποιες εξελίξεις όπου είναι προφανές ότι χρειάζεται βελτίωση σε κάποιους τομείς πολιτικής. Υπάρχουν 27 ε, συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ όλες και όλους τους και οδησηγητές για το έργο τους, ιδίως τον Ίγκορ Σόλτες και τον διαρκή εισηγητή για το Κόσοβο, είναι μάλιστα ο ίδιο και διαρκή εισηγητή για το Κόσοβο. Και για πρώτη φορά έχουμε καταφέρει στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε ταυτόσιμε διατυπώσει και στι δύο εκθέσει και για τη Σερβία και για το Κωσυφοπέδιο. Το θεωρώ αυτό σημαντική πρόοδο, διότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ομιλεί με μια φωνή. Αναμένω τώρα τις παρατηρήσεις σας και βεβαίως και την ε, ψηφοφορία που θα γίνει 8 και 9 Οκτωβρίου. Έχουμε τώρα και ένα εντυπωσιακό κατάλογο εγγεγραμμένων ομιλητών. Μέχρι τώρα είναι 8 συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. 15 λεπτά έχουμε για την συζήτηση αυτή. Παρακαλώ, λοιπόν, δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη και θα βοηθήσει τη Σερβία να κατανοήσει ποιε είναι οι αδυναμίες της και ποια είναι τα ισχυρά σημεία της. Και νομίζω ότι οι χώρε αυτέ θα πρέπει να, από, να να δράξουν αυτή την ιδιαίτερη ευκαιρία που έχουν σε ό,τι αφορά την πρόοδο. Οι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει ω σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν τι σερβικέ αρχέ για κρίσιμα θέματα σε ό,τι αφορά την ενταξία και τη πορεία. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα, το κράτο δικαίου, τη διαδικασία μεταρρύθμισης του δικαίου, τι πολιτικέ ελευθερίε, την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Η Σερβία είναι λοιπόν στην διαδικασία ένταξη ε, και έχει σημειώσει πολύ καλή πρόοδο σε πολλού τομείς, όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη με λειτουργούσα αγορά στις μεταφορές. Είναι σημαντικό ωστόσο να ενθαρρύνουμε, να προωθήσουμε τά αποτελέσματα από τις μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι το δικαστικό σώμα, όπως είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διαφθοράς. Χαιρόμαστε λοιπόν που υπάρχει μεγάλη δέσμευση σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, γιατί η Σερβία είναι ένα εταίρο κλειδί στην όλη περιφερειακή και είμαι πεπισμένο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να του καλωσορίσουμε στην ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία για τη Σερβία και να ακούσουμε τώρα την Τάνια Φαγιόν. Ευχαριστώ, πρόεδρε, και θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω καταρχά για την εξαιρετική συνεργασία μαζί με όλου του κοιόδες. Ιδιαίτερα σε όσα μας αναφέρατε, γιατί όντως υπάρχουν ε, κάποια ευαίσθητα ζητήματα και είναι σημαντικό να έχουμε την ίδια διατύπωση και στις δύο εκθέσεις. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με πολλές από τις συμβιβαστικέ σας λύσεις. Οι τροπολογίες της ομάδας μας συμπεριλήφθησαν σχεδόν όλες στους συμβιβασμού και θα ήθελα ιδιαίτερως να υπογραμμίσω τη συμβαστική υπαριθμό 18 που ενισχύει τα θέματα ελευθερίας του τύπου καθώς και την 21 για τους Ρωμά, τη συμβαστική 21 και χάρηκα που καταδικάσαμε την εκτέλεση του Κωσοβάρου Σερβού πολιτικού στην ε, τροπολογία περιθμών 24. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση και τα μέσα ενημέρωση, παρά το γεγονό ότι αυτό καλύπτεται στη συμβιβαστική τροπολογία και το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο ξανά και ξανά, η κατάσταση στη Σερβία δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να επικρίνουμε τα τεκτενόμενα τα όσα συμβαίνουν στον τύπο και στα μέσα ενημέρωση. εκ παραλλήλου. Δυστυχώ, δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε τις στο Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά τι ε, αρμοδιότητε ε, ελέγχου του Κοινοβουλίου. Και τέλος, η πιο σημαντική τροπολογία, η 25 ε, για τι συνομιλίε μεταξύ Κωσυφοπηδίου και σερβία για την προσαρμογή των συνόρων. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ε, ευαίσθητο και για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και για το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου. Σκοπός μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε την ίδια διατύπωση και στις δύο Το πετύχαμε αυτό, αλλά η εμπειρία μας ε, από τη Σλοβενία ε, μας καταδεικνύει ότι οποιαδήποτε μετακίνηση των συνόρων αποσταθεροποιεί την περιοχή και την περιφέρεια και θα πρέπει να την αποφύγουμε πάσα θεσία. Να υποστηρίξω επίσης τον κύριο Κούκαν για την 133 την τροπολογία. Δεν συμπεριλαμβάνεται στις συμβαστικές. Είναι πολύ σημαντική όμως για το θέμα της κατάχρησης των ε, θέσεων των αξιωματούχων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο θέμα στην ε, Σερβία. Και τέλος, μια προειδοποίηση προς τη Σερβία. Αν δεν προσαρμόσουν την πολιτική τους για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Ιράν μέχρι τέλη Οκτωβρίου, έχουμε λάβει κάποιες ενδείξεις ε, ότι θα είναι αρνητική η έκθεση για το θέμα των θεωρήσεων στα τέλη του χρόνου. Να το λάβουμε λοιπόν υπόψη γιατί είναι σημαντική αυτή η προειδοποίηση προς την Σερβία και στο πώς θα αντιμετωπίζει το όλο θέμα με το Ιράν. Ευχαριστούμε την κυρία Τάγιον, ο Ιβο Βάιγλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και ε, τον Πρόεδρο και εισηγητή και να σας πω πως η έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετική και αποδεικνύει πως η διαδικασία διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στις χώρες που είναι στη νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης. Η Σερβία έχει γίνει ένα κεντρικό κομμάτι αυτής της περιοχής και πρέπει να σας πω πως αυτή η περιοχή ολόκληρη ε, προχωρά προς τη σταθεροποίηση και τις καλέ σχέσει γειτονία. Στην έκθεση τονίζουμε κάποια, αποθέματα, κάποια θέματα οποία είναι ακόμα ε, κάπω προβληματικά. Κράτο δικαίου, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία των μίντια, η αντιμετώπιση των μειονοτήτων και οι επικοδομητικές σχέσεις που θα πρέπει να ε, δημιουργηθούν με όλους τους ενδιαφέρουμενους παίκτες και κυρίως με το Κοινοβούλιο. Η Άλντε είναι αρνητική για την ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Σερβίας Σιφοπεδίου, όπως επίσης και με την οριοθέτηση των συνόρων. Και ξέρετε πως αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης πρέπει να αλλάξει και ο πολιτικός λόγος των ε, Σέρβων πολιτικών όταν αναφέρονται στις γειτονικέ τους χώρες. Οι Σέρβοι, η κυβέρνηση και ο πληθυσμός θα πρέπει να ξέρουν πως θα τους καλοδεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το να εισέλθει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει να αποδεχτεί όλες τις αξίες στις οποίες βασίζεται αυτή, το οποίο σημαίνει και μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ πολύ από τους πράσινους, ο Ίγκο Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ ε, εξαιρετική αυτή η έκθεση και για το κομμάτι που αφορά το Κωσυφοπαίδιο και για τη Σερβία. Και να σας πω πως είναι πραγματικά εξαιρετική η έκθεση. Γιατί, Γιατί συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις τροπολογίες ε, τις οποίες καταθέσαμε, τις οποίες καταφέρατε να συνδυάσετε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς. Και νομίζω ότι περιγράφεται με πολύ ε, σαφή και ακριβή τρόπο την κατάσταση όπως έχει σήμερα στη Σερβία. Πολλές είναι οι καλές πρωτοβουλίες στη χώρα αυτή, σε πολλά σε πολλούς κλάδους. Αλλά υπάρχουν και κάποια κομμάτια που δεν ε, έχουμε την απαραίτητη βελτίωση. Οι συνάδελφοι έχουν ήδη τονίσει ποια είναι τα θέματα αυτά. Κράτος δικαίου, ελευθερία ε, των μίντια, όπως επίσης και τα θέματα μειονοτήτων. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Είναι το ποινικό δίκαιο. Κυρίως τι συμβαίνει με αξιόπινες πράξεις που ε, αφορούν επιχειρήσεις, για παράδειγμα κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, πιστεύω ότι ο, ο ποινικό κώδικας στο σημείο αυτό θα χρειαστεί τροποποίηση. Ε, επίσης, οργανωμένο έγκλημα, πάταξη οργανωμένου εγκλήματος, πάταξη της ε, διαφθοράς. Και εκεί τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα. Πολλά μπορούν να κάνουν και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι πως οι πολιτικοί ανακατεύονται στα θέματα της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Για τις ε, πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη Βουλή και το επίπεδο δημοκρατίας στη χώρα, θέλω να τονίσω πως εκεί δεν είναι σωστό ή Βουλή να χρησιμοποιεί τη διαδικασία του κατεπήγοντος όταν χρειάζεται να εφαρμόσει νομοθεσία δεν θα πρέπει να περνάνε ε, μέσω διαδικασίας κατεπήγοντος ε, τα νομοθετήματα από τη Βουλή. Να σας πω επίσης πως έχουμε ε, διαδικαστικούς κανόνες που καταπατώνται στο, στη Βουλή, γιατί πολλές φορές δεν επιτρέπεται στην αντιπολίτευση να καταθέσει την άποψή της. Και οι σχέσεις γειτονίας μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, ειλικρινά ελπίζω πως επιτέλους στο μέλλον θα δούμε φως μέσα από το τούνελ και θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση και για το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Σόλτε. Φάμπιο Καστάλτο, EFDD. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο ε, Μακάλιστερ για το ότι συμπεριέλαβε πολλές από τις τροπολογίες που καταθέσαμε μέσα σε μια ιστορική στιγμή και θέλουμε να στείλουμε το σωστό μήνυμα στις των Δυτικών Βαλκανίων και να τους πούμε πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάμε μια στιγμή δύσκολη και γι' αυτό ε, θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε και τους άλλους ε, στην περιοχή εκείνη οι οποίοι περνάνε μια διαφορετική στιγμή ιστορικά. Γιατί έχουμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδος, λέει ο και θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τη Σερβία στην διαδικασία προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί. Και το λέει αυτό η έκθεση. Ξέρετε, το πιο ευαίσθητο θέμα είναι η ενδεχόμενη συμφωνία για τα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Ναι, θα πρέπει η διατύπωση σε αυτή τη συμφωνία ε, που θα υπάρχει στη νική Συμφωνία να είναι σωστή, έτσι ώστε να διευκολύνουμε μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να διαχειριστούν με τον σωστό τρόπο και τα δύο κράτη. Γιατί κίνδυνοι εκεί υπάρχουν. Ακόμα. Αλλά η ακινησία των τελευταίων ετών είναι ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι θετικό λοιπόν να δούμε πως αυτή η νέα δυναμική ε, ξεπηδάει στην περιοχή αυτή, αλλά δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από ψευδοενθουσιασμούς Απλώς θέλουμε την ελπίδα πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Η Σερβία είναι βασικό συμμαχός μας στην περιοχή, είναι μια φίλη χώρα και ελπίζουμε πως η Σερβία και οι άλλες χώρες εκείνης της περιοχής κάποια στιγμή θα γίνουν κομμάτι της δικής μας ευρωπαϊκής οικογένειας, παρόλο που ακόμα σήμερα δεν είναι. Ευχαριστούμε τον Φάβιο Καστάλτο και τώρα από την ομάδα του ΙΕΝΕΦ e ο κύριος Σαφχόζε. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα να σας πω πως η Σερβία βεβαίως είναι κομμάτι της Ευρώπης και δεν λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω της Ευρώπης. Euh, Αυτό που θέλω είναι να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όμως σχετικά. Ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Γιατί να το επικρίνουμε η Σερβία έχει ένα ρόλο ουσιαστικό να παίξει. Έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με τη Ρωσία και μπορεί να έχει εξίσου καλέ σχέσεις και με την Ευρώπη. Να είναι γεφυροποιό. και αντί να την επικρίνουμε θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε και να δούμε ποιο είναι ο συγκεκριμένος ρόλος που αναλαμβάνει η Σερβία για να προσφέρει ακριβώ αυτή την ισορροπία. Ξέρω πως οι Γερμανοί προσπαθούν και αυτοί εκεί να πετύχουν μια καλή ισορροπημένη σχέση με τη Ρωσία. Δεύτερον, θα ήθελα στο προήμιο να υπογραμμίσουμε όλα τα σημεία τα οποία είναι σχετικά το ότι ο πόλεμος της δεκαετίας του 90 ήταν παράνομος, πως υπάρχει απόλυτη εθνική κυριαρχία της Σερβίας τότε στο Κωσυφοπέδιο και πως οι θεμελιώδεις ελευθερίες ε, συνδέονται με την εθνική κυριαρχία και μου φαίνεται πως τα στοιχεία αυτά δεν έχουν εμφανιστεί αρκετά στην έκθεση και γι' αυτό έστειλα τις σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακούσαμε πλέον όλους τους κοιόδες εισηγητές και έχω ακόμα επτά συναδέλφους που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Ένα λεπτό έκαστος και ζητώ συγγνώμη. Αλλά έχουμε καθυστερήσει. Η ε, κυρία Ζουίτσα. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ εσάς, τον εισηγητή, για την ε, συνοπτική αυτή και ισορροπημένη έκθεση. Κατέθεσα κάποιες τροπολογίες για σημαντικά θέματα όπως είναι η πολιτική εκπροσώπηση των ε, μειονοτήτων στην Εθνική Εθνοσυνέλευση, στην Εθνοσυνέλευση, στην, τις πολιτικές για την ελεύθερη μετάδοση των μειωτικών γλωσσών στον τύπο και στην τηλεόραση και οι σερβικές αρχές θα πρέπει να επιλύσουν το θέμα των αγνοούμενων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα του πολέμου και τη, τα θέματα διαδοχής ε, της πρώην Γιουκοσλαβία και σε ό,τι αφορά τα θύματα των στρατοπέδων εργασίας. Όλα αυτά τα προβλήματα, Πρόεδρε, θα πρέπει να επιληθούν προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να υποστηρίξουμε τη Σερβία με το παρελθόν της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει και μια εξομάλυνση των σχέσεων με την Πρίστινα και να εκφράσουμε και την πλήρη ε, υποστηρίξη μας για την ε, πορεία της. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στον κύριο Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ. Εξαιρετική είναι η έκθεση για την πρόοδο της Σερβίας τον τελευταίο χρόνο γιατί θεωρώ ότι κάλυψε τα πιο προεξέχοντα θέματα. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόοδο στι διαπραγματεύσει. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα όμω ε, στο κρατό δικαίου, στην ελευθερία του τύπου, σε θέματα δημοκρατία. Κατέθεσα διάφορε τροπολογίε. Θέλουμε να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα Κοιτάξτε, θέλουμε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε πιο πολύ διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών εκστρατιών, των πολιτικών κομμάτων. Όταν μιλάμε για θέματα συνεργασία, λοιπόν, αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη Σερβία, γιατί ενδεχομένω να έχουν και αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν θέματα εκκρεμή οι αγνοούμενοι, η δίωξη των εγκληματιών πολέμου, τα θέματα ιδιοκτησία και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα δε και τις πρόσφατες προτάσεις για ανταλλαγή γεών, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι υπάρχει το πολιτικό πλαίσιο για την εξομάλυνση των πολιτικών σχέσεων και οποιασδήποτε τέτοιε ιδέε ad hoc ενδεχομένω να αποσταθεροποιήσουν όλη την περιφερεια. Να, να παραμείνουμε δηλαδή στο τρέχον πλαίσιο. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο. Ο κ. Επιτίδιο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω κάθε χώρα η οποία επιδιώκει την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και η Σερβία προσπαθεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια τη συνθήκη Κοπεχάγη, και προ αυτή την κατεύθυνση είναι λογικό σε άλλου τομεί να παρουσιάζεται πρόοδο, σε άλλου να υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση προ το παρόν τουλάχιστον. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη Σερβία με μια προκατάληψη. Πρέπει να την αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει και τι υπόλοιπε χώρε των Δυτικών ε, Βαλκανίων που επιδιώκουν ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κρίνεται η πρόοδο σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με βάση την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνονται. Δεν μπορεί να αποτελέσει και δεν πρέπει να αποτελέσει η προσπάθεια της Σερβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντικείμενο εκβιασμού τη χώρα αυτή να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική και να αρνηθεί την εθνική τη κυριαρχία. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα αναταραχή στα Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε. Και να εμείνω σε κάτι πολιτικό, όχι για τη Σερβία, αλλά για την επιρροή στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Γιατί σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε εκλογές και έχουμε απευθύνει ε, έκκληση προς τον κύριο Βούτιτς για να ε, μετριάσει τις αντιδράσεις τους και σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα είπε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το θέμα του Ντόντι. Τώρα υποστηρίζει όμως τον Ντόντι σε μια προεκλογική εκστρατεία που επικρίνει τη δυτική επιρροή στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ένα πολιτικό λοιπόν παράγοντα λοιπόν στην, στην ε, περιοχή, στην χώρα που πρόσκειται στον ε, Πούτιν και υποστηρίζει τον πρόεδρο Βούτσης ε, κατά της δύση. Ε, νομίζω ότι η Βοσνία θα έπρεπε να στραφεί προς την ευρωπαϊκή πορεία, όχι να ακολουθήσει την πορεία της Μόσχας, της Μόσχας στην φτωχή χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ως μέλος της αντιπροσωπεία στη Σερβία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την πολύ καλή έκθεση. Και νομίζω ότι θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση τη συζήτηση μα όταν θα επισκεφτούμε το Βελιγράδι τέλη Οκτωβρίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όλου ιδιαίτερω αυτό που αναφέρετε στην έκθεσή σα για το κράτο δικαίου και πόσο σημαντικό είναι να καλωσορίσω και την αναφορά στο θέμα της πρόσβασης ε, στην δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά και το άρθρο 47 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ξέρω ότι σημείωσατε πρόοδο στου συμβιβασμού, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε τελική ανάλυση πιστεύω όσο πιο πολλοί συνάδελφοι να υποστηρίξουν την περαιτέρω πρόοδο για την ε, επικέντρωση στον κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική συνεργασία, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα προωθήσει τις ευκαιρίες της Σερβίας για την ε, ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ζωφκό. Να σας συγχαρώ και εγώ για την πολύ καλή αυτή έκθεση, καθώς και για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στην ευρωπαϊκή πορεία της. Οι τροπολογίες μου, παρά το γεγονός ότι δεν έχω ακόμα εξετάσει τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και έτσι δεν μπορώ να αποφανθώ επ' αυτών, οι δικές μου τροπολογίες αφορούν τη μετανάστευση, την απελευθέρωση του καθεστώτος ε, θεωρήσεων με το Ιράν, και τη διευκόλυνση της απελευθέρωσης από το καθεστώς θεωρήσεων με άλλες χώρες. Επεσήμενα ότι η Σερβία θα πρέπει να εξετάσει την πολιτική αυτή. Γιατί ενδεχομένω να έχει συνέπειε και σε χώρε που δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βοσνία Ζεγοβίνη, όπου καταφτάνουν σε κύματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταχρώμενοι της κατάστασης ε, με σκοπό φυσικά να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα για την Κροατία που έχει το μεγαλύτερο σύνορο με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Σερβία λοιπόν θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της διακίνησης μεταναστών γιατί πρόκειται για μια επικερδή μπίζνα η οποία επιβαρύνει την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ζαφκό και τέλος η κυρία Άλιου Μαρή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να πω τίποτε για την έκθεση ούτε για το Κόσοβο. Έχω μια ερώτηση ωστόσο. Στις εκθέσεις αυτές για τις υποψήφιες χώρες, υποψήφιες για ένταξη, γιατί δεν διαβάζουμε ποτέ τίποτε σχετικά με τις πρόοδους που μπορούν να επιτευχθούν υπέρ των πολιτών των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόοδο και το επίπεδο ευημερία. Θεωρώ, το βιωτικό επίπεδο δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μόνο για να αναπτύσσει τις οικονομίες, ασφαλώς και για να φροντίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά μέσα στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών των χωρών αυτών δεν πρέπει να προβλέπεται και η βελτίωση της οικονομική του ευμάρεια. Μέσα στις εκθέσει αυτέ δεν μιλούμε ποτέ για τα πράγματα αυτά. Αν θέλουμε μια πραγματική ενότητα, αν θέλουμε πραγματικά να ξυπνήσουμε στου πολίτε αυτού το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια Ενωμένη Ευρώπη, πρέπει να του δείξουμε κιόλα ότι η Ενωμένη Ευρώπη βελτιώνει την καθημερινή ζωή του καθενό, επομένω και την ηλική του ευζοία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να περνάει σε όλε τι εκθέσει αυτέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία άλλη Μαρή είναι ε, ισχυρό το επιχείρημά σας, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν πολύ τεχνικό χαρακτήρα και ίσως στην γλώσσα που χρησιμοποιούμε να μην καλύπτουμε 100% όλα τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Πολύ σωστό λοιπόν το θέμα που θίγεται και ίσως μπορούμε να το βάλουμε την επόμενη φορά. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις σας ψηφοφορία στις 9 Οκτωβρίου, εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών. Το υπαριθμόν 7. Έκθεση για την έκθεση της Επιτροπής 2018 για το Κωσυφοπέδιο ή Κόσοβο. Τον λόγο λαμβάνει ο εισηγητής Ίγκορ Σόλτες. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ειλικρινώς επίσης όλους τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι θεωρώ ότι έδειξαν μεγάλη διαθεσιμότητα και προθυμία να δεχτούν και τις τροπολογίες που συντάξαμε. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία βεβαίως, καθώς και τους συμβούλους οι οποίοι ε, συνέβαλαν στην ε, σύνταξη των συμβιβαστικών τροπολογιών, οι οποίες συμβαστικές τροπολογίες περιλαμβάνουν και κάποια από τα κέρια μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Κόσοβο. Στο παρελθόν, πέρσι μάλλον πιο συγκεκριμένα, μετά δηλαδή από την ψήφιση της ε, τελευταίας εκθέσεως, έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα και θα ήθελα να φωτίσω ιδίω το ζήτημα της απελευθέρωσης των προξενικών θεωρήσεων. Ως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το Κόσοβο πληρεί πλέον τους όρους και θεωρεί ότι το Κόσοβο, η Κωσυφοπαίδιο, θα πρέπει να λάβει το πράσινο φω για την απελευθέρωση του καθεστώτος προξενικών θεωρήσεων. Στην τελευταία του ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση έδωσε το πράσινο φω για την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσουμε τώρα από το Συμβούλιο Υπουργών να κάνει και αυτό το αναγκαίο βήμα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα, διότι θα βοηθήσει να αποκατασταθεί μια ισορροπία και μια ισότητα στην περιοχή αυτή. Θα μας επιτρέψει επίσης να περιλάβουμε το κοσυφοπεδίο σε όλες τις διαδικασίες που εξελίσσονται στην περιοχή αυτή και που όλες θα έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στους διαφόρους άλλους τομείς. Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει και την πρόοδο που έχει γίνει στα διάφορα θέματα, αλλά και θέματα τα οποία πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη του, οι αρχέ του κοσυφοπεδίου. Οι όροι για την απελευθέρωση του καθεστώτο των μοξενικών θεωρήσεων θεωρούμε ότι πληρούνται. Από την άλλη μεριά όμως οι αρχέ του Κωσόβου πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθορά. Θα χρειαστεί λοιπόν να ιδρυθεί ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς Επίσης ζητήματα ασύλου πρέπει να επιληθούν. Το Κόσοβο καλείται να παίξει ρόλο σε όλες τις διαδικασίες του μεταναστευτικού και γι' αυτό το Κόσοβο θα πρέπει να καταδείξει ότι εφαρμόζει μια αποφασιστική πολιτική στην, ε, στην υπόθεση αυτή. Γνωρίζετε ότι ε, δολοφονήθηκε ο Ιβάνοβιτς και θέλουμε να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος αυτού. Τονίζω ένα άλλο σημαντικό θέμα, τον ρόλο δηλαδή των γυναικών στην ε, κοινωνία του Κωσόβου, καθώς επίσης και την στάση απέναντι σε μειονότητες, απέναντι σε αναπήρους, διότι σε όλους αυτούς τους τομείς απαιτείται πολύ και εντατική εργασία από τις αρχές του Κωσυχοπεδιού. Εν τέλει, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο ακόμη σημαντικά θέματα. Πρώτο, το Κόσοβο και η Σερβία οφείλουν πλέον να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των και να βελτιώσουν τις σχέσεις των. Χρειαζόμαστε οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ άλλων στον αθλητισμό και πιστεύω ότι αν δώσουμε πράσινο φως σε έργα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις των δύο χωρών, όπως για παράδειγμα στον αθλητισμό, αυτό θα βελτιώσει και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τέλος, περιβάλλον. Η Πρίστινα είναι από τις πόλεις εκείνες που ε, θίγονται βαρύτατα στην περιοχή αυτή από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ζητούμε από τις αρχές λοιπόν να φροντίσει να κάνει πολύ περισσότερα για να βελτιώσει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και επομένως και τη ζωή των πολιτών της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ίγκορ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πρώτα στον Τονίνο Πίτσολα που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας με την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω το εξή. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Γιατί λαμβάνει υπόψη και τη, διάσκεψη, τη διάσταση του κοσυφοπεδίου και αναφέρεται σε όλα τα όσα συνέβησαν πέρυσι. Είμαι πρόεδρος ή μάλλον επικεφαλής της αντιπροσωπείας και θα ήθελα να τονίσω το εξής. Πήγαμε στην Πρίστινα την περασμένη εβδομάδα και ήταν η πέμπτη συνάντηση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Κωσυφοπαίδιο. Και αντίθετα με τόσο συνέβηνα όταν συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο και μετά από κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε στην αρχή, πρέπει να σας πω πως τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, καταλήξαμε σε συμπεράσματα και συστάσεις όταν τελείωσε η συνάντησή μας. Και πρέπει να σας πω ότι μεν πέρσι έγιναν πολλά, Είχαμε και τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απελευθέρωση της χορήγησης θεωρήσεων και ελπίζω πως όλα αυτά σύντομα θα κλείσουν και οι πολίτες του κοσφοπεδίου θα μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους επιτέλους να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πολλά μένουν για τη μάχη κατά της διαφθοράς, για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης και για την εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν στα πλαίσια του διαλόγου με τη Σερβία. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται μια συμφωνία γενική μεταξύ Σερβίας και Κοσφοπεδίου που θα πρέπει να επιτρέπει στα δύο αυτά κράτη να ε, συμφωνήσουν κάτι χωρίς αυτή η συμφωνία να έχει αρνητικές συνέπειες είτε στο εσωτερικό των δύο χωρών είτε στην ευρύτερη περιοχή. Σκιώδεις εισηγητές τώρα. Ε, να ξεκινήσουμε με το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πήγα σε αυτή την πέμπτη συνάντηση ε, στο Κωσυφοπέδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να τους πω ότι χαίρομαι που έχουν ε, συμμορφωθεί με τους κανόνες για την απελευθέρωση ε, των θεωρήσεων, την απαλλαγή μάλλον από την υποχρέωση θεωρήσεων, όπως μας είπε τον Ιούλιο Κομισιόν και όπως αποφασίσαμε στο Στρασβούργο. Χαίρομαι που έχει ε, σημειωθεί πρόοδο. Χαίρομαι που έχουν προχωρήσει οι οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο και χαίρομαι που ανοίγεται μια προοπτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κεντρικό σημείο και το πιο κομβικό είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Σερβίας και Κοσφοπεδίου. Πολλά έχουν ακουστεί. Εμείς στηρίξαμε απόλυτα τη συνέχιση του διαλόγου, όπως επίσης και την ενδεχόμενη ε, εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας. Όλοι θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να τους βοηθήσουμε να εξομαλυνθούν οι σχέσει του γιατί αυτό αποτελεί και μία από τι σχέσει για τι δύο χώρε και για τη Σερβία και για το Κωσυφοπέδιο, για να μπορέσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται βέβαια πρόοδο, διαφθορά, κράτος δικαίου, αλλά είμαι χαρούμενη που έχουν εγκρίνει πρόσφατα νόμου για την καταπολέμηση τη διαφορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Ευχαριστώ, Ιγκορ Σόλτε. Ευχαριστώ για την πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Από σοσιαλιστές, ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδεις γιατί είναι μια σημαντική στιγμή η χρονική στιγμή που διανύουμε. Είναι ισορροπημένο το κείμενο και περιγράφει καλά την κατάσταση στη χώρα και δείχνει και ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι επιτυχίες και τι θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση του δημοσίου, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, πάταξη της εγκληματικότητας, της διαφθοράς. Όπως είπατε και εσείς, το κοσυφοπέδιο επιτέλους πληρεί ε, τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων και θα το αποφασίσει αυτά το Συμβούλιο και ελπίζω με τον τρόπο αυτό θα ευνοηθεί και η διαδικασία σταθεροποίησης και συνεργασίας σε αυτή την γεωγραφική ζώνη που είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Κωσυφοπεδίου-Σερβίας, καλό θα ήταν οι πέντε χώρες που ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο να το κάνουν. Και να υπογραμμίσουμε πως ο ορισμός και η χάραξη των και η οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κοσμοπεδίου θα πρέπει να γίνει μέσω διαλόγου και συμφωνίας και όχι να βασίζεται μόνο σε εθνοτικά κριτήρια. Τώρα για τις πολιτικές, για το, για το φύλλο, για τις μειονότητες, για τις διακρίσεις, για τους λόάδ ελπίζω πως αυτά θα γίνουν εκεί έτσι ώστε να διευκολυνθεί μέχρι το 2025 η διαδικασία ένταξης. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παντζέρη. Από την άλλη τώρα ο κύριος Ράμος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματο τη συναδέλφου Γιλντε Λάιτμαν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτα για την εξαιρετική συνεργασία. Και που έλαβε υπόψη διάφορε τροπολογίε που κατέθεσαν και οι συνάδελφοι της Άλντα και άλλες πολιτικές ομάδες και που θεωρώ ότι συμπλήρωσαν την ε, έκθεση. Το κοσυφοπέδιο τα συνηθισμένα προβλήματα αντιμετωπίζει όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Όλες είναι αντιμέτωπες ε, με παρόμοια προβλήματα πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, θέματα δικαιοσύνη, διαφθορά, ε, οργανωμένου εγκλήματο. Το Κωσυφοπέδιο, ωστόσο, αντιμετωπίζει και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Το θέμα τη συμφωνία με τη Σερβία, η οποία πρέπει να συναυθεί και θα πρέπει να ενσωματωθούν και οι Σέρβοι όπου αποτελούν πλειοψηφία στο σύστημα, υπήρξαν κάποιες ε, θετικέ ε, ενδείξει η επικύρωση της συμφωνίας με το Μαυροβούνιο, κάποιοι νόμοι, κάποια νομοσχέδια που πέρασαν σε ό,τι αφορά και τις προδιαγραφέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα του δικαστικού και το θέμα α, ε, της Βόρειας Σερβίας και της ένταξης των εκπροσώπων αυτών στο δικαστικό σύστημα. Μιλάμε για τεράστια λοιπόν βήματα στο κοσμοπέδιο. Το κοσμοπέδιο προφανώς και είναι ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνε του αλλά προφανώς και να ασκήσει και τα δικαιώματα του ως ανεξάρτητο κράτος. Θα πρέπει να δραματίσει και το ρόλο που του αναλογεί στο διεθνές προσκήνιο. Θα πρέπει όλες αυτές οι εξελίξεις να επιταχυνθούν προκειμένου να μπορέσει το κοσμοπέδιο να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες χώρες στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Καστάλντο από το EFTD για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ίγκορ Σόλτες για την εξαιρετική δουλειά που κάνει και για το γεγονός ότι συμπεριέλαβε σχεδόν όλες τις τροπολογίες μου στο κείμενο. Νομίζω ότι ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, σήμερα ε, θα βοηθήσουν το κοσυφοπαίδιο να ευαισθητοποιηθεί και να κάνει ό,τι χρειάζεται μέσω των διαδικασιών και των κοινοβουλευτικών εκεί που θα τους βοηθήσει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν μεταρρυθμίσεις, προεκλογικό σύστημα, διαφθορά, κράτος δικαίου. Πάρα πολλά χρειάζονται να αναμορφωθούν και ελπίζω πως η Βουλή τους θα μπορέσει να τα αναλάβει με πιο ταχύς ε, ρυθμούς. Θα πρέπει η απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων να είναι ένα κίνητρο. Το κοσφοπέδιο σήμερα αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά έχει και μεγάλες ευκαιρίες και δεν θα πρέπει να τις αφήγουν να ξεφύγουν εταίρων. Λοιπόν, με τη Σερβία θα πρέπει να βασίζονται σε μια συνεργασία πραγματική. Να έχουν επαφή μεταξύ των εθνών, να υπάρχει διάλογος και όπως έχουμε πει για την ε, Σερβία, η ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ της Σερβίας και του Κουσουβοπαιδίου είναι μία από τις καλύτερες δυνατές πιθανές εξελίξεις. Και νομίζω ότι το κείμενο θα πρέπει να είναι ίδιο και στις δύο εκθέσεις. Γιατί αν δεν αλλάξει η δυναμική θα παραμείνει σε αυτή την ε, κατάσταση το κοσυφοπαίδιο σε ένα είδος, ε, σε μια ασάφεια θολή ε, νομικά, κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά θα πρέπει να ανασκουμποθούν να προσπαθήσουν και τη δική μας, τις δικές μας επικρίσεις να τις λάβουν ως επικοδομητική ε, προσπάθεια ε, βελτίωσης, στήριξης με συγκεκριμένε αποκρίσεις που θα μας δώσουν και που θα στείλουμε κι εμείς, γιατί θέλουμε σύντομα και αυτοί να γίνουν κομμάτι της οικογένειές μας. Ευχαριστούμε για τους μη κεκραμένους να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σνόσνικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα θέμα το οποίο οφείλεται στην ανεύθυνη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κωσυφοπέδιο. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρατάσσεται με προσώπους της Σερβίας και αυτό είναι απαράδεκτο. Εφόσον έχει το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως που είναι δικαίωμα, αν έχει λοιπόν το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεω, τότε πρέπει να έχουν, έχουν δηλαδή οι κάτοικοι του Κωσόβου, πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα και οι Σέρβοι κάτοικοι του Κωσόβου. Ορισμένοι Σέρβοι δεν θέλουν να κατοικούν στο Κόσοβο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Γιατί δεν γίνεται σεβαστό και γιατί εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά στο ίδιο θέμα. Εφόσον μιλούμε για δικαίωμα αυτοδιαθέσεως, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο πάντα, ούτε θεωρώ ότι ο εθνικισμός πρέπει να είναι η βάση για τη δημιουργία κράτους, αλλά γιατί δεν ισχύει το ίδιο δικαίωμα αυτοδιαθέσεως για όλους εκεί, εκεί όπου υπάρχει για παράδειγμα μια πλειοψηφία Σέρβων και δεν θέλουν να ανήκουν στο Κόσοβο. Γιατί αναγκάζονται οι Σέρβοι αυτοί να είναι πολίτες ενός αλβανικού κράτους ενώ δεν θέλουν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστά τα μέτρα και σταθμά αυτά. Εφόσον όμως τα χρησιμοποιούμε, ας χρησιμοποιούνται προς πάσαν κατεύθυνση. Okay, thank you. Πρόεδρος Μακάλιστερ, ευχαριστώ. Τώρα, μένουν τρεις ακόμη ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Κούκαν, Ward και μετά ο κύριο επιτήριο. Άλλο κανείς? Όχι. Ωραία. Κλείνω τον κατάλογο λοιπόν εδώ. Ο Κούκαν πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την καλή δουλειά που έκανε. Χαίρομαι και για το αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας στην Ολομέλεια για τις προξενικές θεωρήσεις του Κωσόβου και ελπίζω και το Συμβούλιο τους επόμενους μήνες να κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Είναι πολύ ταραγμένη η περιοχή του Κωσόβου και νομίζω ότι πρέπει να το απηχούν αυτό αντικειμενικά οι, οι ε, εκθέσεις. Η διακομματική συνεργασία είναι σημαντική, διότι χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στο Κωσόβο Και αυτό θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκό μέλλον του Κωσόβου. Διότι οι πολίτες του Κωσόβου πρέπει να δουν πραγματικές απτές πρόοδους. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που παραμένουν ακόμη, όπως η βελτίωση Τη κοινοβουλευτικής διαδικασία, όπως λέει η έκθεση και που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Ο διάλογος μεταξύ Πριστίνας και Βελιγραδιού πρέπει να ληφθεί υπόψη με πιο σοβαρό τρόπο και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να δώσουμε δε υποστήριξη και στο Κόσμο και στη Σερβία στη διαδικασία αυτή. Εν τέλει, συγχαίρω τους ηγέτες του Κωσόβου για τη συνεργασία τους με άλλες πλευρές και την ε, ε, ευθυγράμμισή τους με την ε, εξωτερική μας πολιτική. Ευχαριστώ, Κούκαν, η κυρία, η κυρία Ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Είμαι μεγάλη φίλη του Κωσόβου και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει μόνο τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών να εκφράζουν άποψη για το πού θα πρέπει να πάει το Κόσοβο. Εγώ είμαι μέλος ε, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών αλλά και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Και αυτά τα πράγματα με απασχολούν πολύ και στην περίπτωση του Κωσόβου. Ε, είμαι και μέλος στην αντιπροσωπεία ε, για συνεργασία με το Κόσοβο και χαίρομαι πολύ για την δουλειά που έκανε ο κύριος Σπίτσουλα και τον συγχαίρω για τον τρόπο με τον οποίο γύρθηκε τη αντιπροσωπεία την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπορέσαμε να κρατήσουμε το Κόσοβο παρόλο που ορισμένε φορές πέρασε από περιόδου μεγάλη αστάθειας. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Κόσοβο για να του δούμε, έρχονται τα πρόσωπα αυτά και ε, μας βλέπουν και αυτοί και, βρίσκουμε πάντοτε ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Και αυτό είναι σημαντικό για όλα τα Βαλκάνια. Οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου έχουν περιμένει μακρότατο χρονικό διάστημα και ιδίω οι νέοι έχουν περάσει μέσα από πολλέ ταραχέ και αστάθεια και είναι σημαντικό για αυτούς να ανοίξει μια πορεία προς τα εμπρός. Οι νέοι του κοσυφοπεδίου αισθάνονται Ευρωπαίοι. Ήδη αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και νομίζω ότι πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα να ασκήσουν και όλα αυτά δικαιώματα αυτά δηλαδή. Και ο κ. Σόλτες και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω να συνεχίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρόοδο ε, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και του Κωσυβεποδίου πρέπει να κριθεί αντικειμενικά με βάση των επιδόσεων της χώρας αυτής. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται να διανύσει μεγάλο δρόμο ακόμη για να έχει θετικέ ε, προοπτικές. Ξέρουμε ότι το Κόσοβο είναι μία από τι πλέον διεφθαρμένε χώρε της Ευρώπης. Επιπλέον υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και έχει αποτελέσει η χώρα αυτή καταφύγιο πολλών τρομοκρατών φανατικών τζιχαντιστών. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία και ευαισθησία έχουν οι πολιτικές επιλογές του Κωσυφοπεδίου. Πρέπει να χαραχθούν τα σύνορα με το Μαυροβούνιο, με τη Σερβία και εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να προσεχθεί είναι η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου να ομοσπονδιοποιηθεί με ένα άλλο κράτο το οποίο επιδιώκει την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλβανία. Όπω ξέρετε, η αλβανική κυβέρνηση, αν δεν υποστηρίζει, στην καλύτερη περίπτωση ανέχεται κάποιε επεκτατικέ βλέψει ορισμένων οργανωμένων ομάδων. Άρα λοιπόν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ε, ε, ασφάλεια αλλά και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Τέλο, αυτή ακριβώ η κατάσταση με το γεγονό της δημιουργίας de facto αυτού του κράτους αποτελούν και τους βασικούς λόγους για τους οποίους ορισμένα κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα δεν έχουν αναγνωρίσει τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επιτίδη. Δεν έχω άλλα σχόλια, άλλες παρεμβάσεις. Σας ενημερώνω ότι η ψήφος ε, θα λάβει χώρα 9 Οκτωβρίου και προχωρώ στο υπαριθμό 8 με μισή ώρα καθυστέρηση βεβαίως σημειώνω πρόκειται για την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της ΑΦΕΤ σε Τινησία και Αλγερία ελπίζω ότι θα χρειαστεί κάπως λιγότερος χρόνος από αυτόν που έχουμε προβλέψει για την συζήτηση αυτή λοιπόν αποστολή της ΑΦΕΤ πήγε στις δύο αυτές χώρες, την Ισία Αλγερία, από 16 έως 20 Ιουλίου, εβδόμου δηλαδή, πρώτα 16 με 18 στην Ισία, με επικεφαλής τον κύριο Γιώ Λάινεν, τον οποίο καλωσορίζω εδώ, και ανάποδα μάλλον, η Αλγερία πρώτη. Και έγινε η συνάντηση στην Τινησία για ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων εκεί. Θα τα ακούσουμε αυτά από τον Γιό Λάινεν. Πριν όμως του δώσω τον λόγο, να σας πω δύο λόγια για το δεύτερο μέρος της αποστολής, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πήγε η αποστολή και στην Αλγερία. Και λίγους, ε, λίγες εβδομάδες μόνο μετά από την ίδρυση της σχετικής αντιπροσωπείας για να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και την κοινοβουλευτική συνεργασία με την Δημοκρατία της Αλγερίας. Καρποφόρες συναντήσεις με Πρωθυπουργό, η Υπουργό Εσωτερικών και άλλους υψηλούς αξιωματούχους. Ήταν ε, ανοιχτές και γόνιμες οι συζητήσεις για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ε, Αλγερίας, καθώς και για την ασφάλεια της περιοχής. Ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής, η Αλγερία παίζει σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο και είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί η συνεργασία για θέματα ασφαλείας, καταπολέμηση τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποίηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Γιώ Λάινεν για την Τινησία. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Φρόντισε με θαυμάσιο τρόπο να προετοιμάσει την αντιπροσωπεία η Γραμματεία και την ευχαριστώ πολύ. Στην Τινησία είναι ασταθής η πολιτική κατάσταση. Μόλις στην Προτεραία είχε δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση ο πρόεδρος και είχε αμφισβητήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι του χρόνου θα γίνουν κοινοβουλευτικές εκλογές και ήδη τοποθετούνται τα κόμματα σχετικά. Ξέσπασε λοιπόν πραγματική πολιτική θύελα, δεν μπορέσαμε να δούμε λοιπόν ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τον Υπουργό Ιστορικών. Είδαμε όμω ε, άλλα ε, πρόσωπα στο Κοινοβούλιο, δηλαδή βουλευτέ, αλλά και εκπροσώπους της ε, ε, Κοινωνία των πολιτών και ιδίω εκεί μα απασχόλησε η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων από πέντε θεσμούς που έχουν υποσχεθεί να ιδρύσουν μόνο η Επιτροπή Εκλογών. Δεν υπάρχει ούτε ακόμα συνταγματικό δικαστήριο, δεν έχει γίνει μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου, ούτε του συστήματος ασφαλεία μας παραπονέθηκαν για ε, εκτεταμένη και παρατεταμένη ατιμορρησία, διότι το σύστημα δικαιοσύνης δεν λειτουργεί. Διαπιστώσαμε και μια απογοήτευση των νέων με 30% ανεργία, παρακαλώ, ε, κακό εκπαιδευτικό σύστημα. Η Τινησία είναι μια νεαρά χώρα και πολύ νεαροί Τινήσοι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι διότι δεν βλέπουν μέλλον. Αυτό ε, οφείλεται και σε μια στατικότητα της οικονομίας και στασιμότητα συγγνώμη, της οικονομίας. Ε, λίγες οικογένειες ε, χειρίζονται τα της οικονομίας και δεν κινείται τίποτα εκεί. Υπάρχει για παράδειγμα ένα μονοπόλιο ενέργειας όπου οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου διότι ε, το ενεργειακό μονοπόλιο είναι μια χαρά ευχαριστημένο με την ενέργεια που διαθέτει και πολύ του χρόνου γίνονται κοινοβουλευτικές εκλογές, όμως τον Μάιο έγιναν δημοτικές εκλογές με επιτυχία. Οι δημοτικές εκλογές δηλαδή πέρασαν το τεστ, ας πούμε έτσι, για πρώτη φορά υπάρχουν περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια και ε, θα είναι σημαντικό τώρα, τώρα να εφαρμοστεί όντως η αποκέντρωση με τη χορήγηση αρμοδιοτήτων αλλά και χρηματοδότησης στα, στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, διότι δεν επιτρέπεται να μείνουν χωρίς καμία στήριξη. Μιλήσαμε βέβαια και για τη μετανάστευση. Η Τινησία είναι και χώρα εισαγωγή μεταναστών από την υποσαχάρη Αφρική, αλλά και ε, χώρα ε, διάβασης των μεταναστών και μας είπαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να φτιάξουν ε, κέντρα υποδοχής μεταναστών. Ωστόσο, για ζητήματα συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Αμήνης μας μίλησε και για την ασφάλεια, είπε ότι υπάρχει τρομοκρατία και στα σύνορα προς την Αλγερία, μάλιστα προ λίγου είχε γίνει, λίγες ημέρες πριν από, την, από το ταξίδι μας εκεί, είχε γίνει ε, σχετική ε, τρομοκρατική επίθεση, αλλά και στα σύνορα προς την Λιβύη φτωχή χώρα την Ισία, ωστόσο δίνει 15% του προπολογισμού της για ζητήματα άμυνας. 15% είναι πολλά χρήματα. Εν τέλει, ε, συναντηθήκαμε και με την Επιτροπή Αληθείας και Αξιοπρεπίας. Υπάρχουν 50.000 προσφυγές ενώπιον της Επιτροπής αυτής για ζητήματα προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήδη από την ε, εποχή του Προέδρου Αλή, Μπεν Αλή. Δεν παρατάθηκε ωστόσο η εντολή της ε, ε, επιτροπής αυτής που θα ήταν σωστό διότι έρχονται τώρα κάποιες πολύ σημαντικέ υποθέσεις και είδαμε ότι αυτή η θαυμάσια Επιτροπή με δική τη πρωτοβουλία αλλά και με δική τη ανάληψη κόστους επιθυμεί να συνεχίσει μέχρι τέλου του έτους. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο συμφέρον να στηρίξει την ε, δημοκρατική και οικονομική πορεία τη Τινησία, και θα χρειαστεί ε, να εγγύψουμε πάρα πολύ προσεκτικά στην ε, κατάσταση στη χώρα αυτή. Σα ευχαριστώ Γιώλα, Λάινεν, λέει ο Ντέβιν ε, Μακάλιστερ για την τοποθέτησή σας. Έχουμε τώρα δύο ε, ομιλητές, Μιλάν Μον και Λόπεθ. Εσείς κύριε Μιλάν Μον. Δεν είχα ζητήσει το λόγο μου, αλλά αφού μου τη δίνετε, να την πάρω την ευκαιρία αυτή και να σας πω ότι δεν έχω να προσθέσω και κάτι το ιδιαίτερο. Είναι σημαντικό πάντως να δούμε το θέμα των ε, πολιτικών μεταρρυθμίσεων και να δούμε τι γίνεται και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, γιατί εκεί μεταρρυθμίσεις πολλές δεν έχουμε. Και είναι ένα αρτήριο σκληριωμένο κράτος σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει μια έλλειψη ενθουσιασμού στην νεολαία και δεν υπάρχει αυτό το boom το οικονομικό και το κοινωνικό στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν γιατί υπάρχει πάρα πολλή ενεργεία και γιατί είναι ε, μια περιοχή που, από που όχι μόνο περνάνε μετανάστες αλλά φεύγουν και πάρα πολλοί νέοι. Και φεύγουν για Ιταλία, για οπουδήποτε. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια χώρα όπου οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις δεν ξεκίνησαν στο, τουλάχιστον όχι με αρκετά με αρκετή θέρμη και να σας πω πως ο υπουργό Άμυνας παραπονιέται πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μας ζητάνε να τους λύσουμε τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και αυτοί για να τους βοηθήσουμε πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, να μην περιμένουν όλα να τα κάνουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κ. Λόπες. Muchas gracias, presidente. Ε, Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να πάρω το λόγο και να σας πω πως οι επισκέψεις μας πήγαν καλά ένα. Ένα έχω να τονίσω, το πόσο σωστό ήταν που πήγαμε σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι περιοχές που είναι πολύ σημαντικές για μας είναι η Βόρειο Αφρική. Εκεί έχουμε το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, ε, τις και εκεί έχουμε πολύ καλές σχέσεις και πάμε πολύ συχνά. Να σας πω πως για την Τινησία είναι μια χώρα που εμείς το εξωτερικό θεωρούμε πως αποτελεί τη μοναδική επιτυχία των πολιτικών ε, γεγονότων ε, της Αραβικής Άναξης πριν από μερικά χρόνια, αλλά παρόλα αυτά σε εσωτερικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ασταθής και το πολιτικό της σύστημα ε, μοιάζει, αν το πω ανοιχτά, εύθραυστο. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αστάθειας οδηγεί και σε μία εξάντληση γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν πήγαν καλά, χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες και αυτό αποτελεί και κομμάτι των διαμαρτυριών που είχαμε τότε στον αραβικό κόσμο. Οπότε προσέξτε, είναι μια χώρα που, στηρίζει, που χρειάζεται στήριξη. Τώρα η Αλγερία είναι ένα πολιτικό σύστημα που είναι πάρα πολύ τραυματισμένο από την, τον εμφύλιο της δεκαετίας του 90. Είναι μια χώρα που έχει απεικιοκρατικό ε, παρελθόν. Είναι μια χώρα κλειστή, αδιαφανής ε, φοβία, Ισλαμισμός, ερμητικά κλειστή, εσωτερικό κενό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε τους πόρους, έχουμε τη σταθερότητα στην περιοχή, έχουμε τη μετανάστευση και τέτοιου είδους ε, αποστολές βοηθούν και μας υποδέχτηκαν, πρέπει να πω τουλάχιστον στην Αλγερία, σε πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο. Thank have... ευχαριστώ και τώρα έχουμε δύο ακόμα μελητές. Τον Φάμπιο Καστάλδο και τον κύριο Σόσνιετς. Και μετά κλείνει ο τον των ομιλητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, David. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι έγινε αυτή η αποστολή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί θα ξέρετε ότι εξετάζω και παρακολουθώ στενά τι εσωτερικέ εξελίξει στι δύο αυτέ χώρε. Ήμουν άλλωστε και εισηγητή ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τινησία και έχω μεταβεί διάφορες φορές στην αποστολή παρατηρήσεις των εκλογών. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση. Και ίσως με τον τρόπο αυτό μάθουμε και επιπλέον στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην μελλοντική μας αποστολή. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση σε ό,τι αφορά α, την ισορροπία, την κυβερνητική που έχει σχηματιστεί στη χώρα, η οποία είναι υποκατάρρευση. Και αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει στη τελική ανάλυση την σύγκρουση μεταξύ Προέδρου και Πρωθυπουργού. Και αυτό προφανώς οδηγεί στον κίνδυνο συνταγματικών ε, περιπλοκών για θέματα τα οποία ακόμα δεν ε, έχει ρυθμίσει το συνταγματικό δικαστήριο. Και είναι προφανής η σύγκριση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων που σε τελική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα στη χώρα σε ό,τι αφορά την σε εκλογέ. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σα απευθύνω αγαπητοί συνάδελφοι είναι το εξή, Έχετε την εντύπωση ότι αυτές οι εντάσει, αυτές οι τερβέ θα δυσκολέψουν την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεων που είναι πραγματικά κατεπίγουσες για την υπέρβαση των προβλημάτων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αν δεν λάβουν λοιπόν υπόψη, αν δεν λάβουν χώρα αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αυτό ενδεχομένω να αλωτριώσει τους ε, νέους ιδιαίτερους από την ε, τρέχουσα κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας ε, άποψη. Πώς εκτιμάτε την ε, πολιτική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες ε, μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζόσνετς, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για αυτή την αποστολή. Να σα πω πω καταρχήν δεν ήταν καλή ιδέα να πάμε και στι δύο χώρε σε μία αποστολή, γιατί χρειάστηκε να βιαστούμε. Και δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα, σε πολλέ περιπτώσει να κάνουμε τι συναντήσει μα με την ησυχία μα. Και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να μιλήσω για το τι γίνεται με τις εκκλησίες που κλείνουν. Και με ρώτησαν ε, εκπρόσωποι της χριστιανικής κοινότητας στη χώρα μου και δεν είχα μία απάντηση να τους δώσω. Επίσης, η τεράστια διαφορά στην προσέγγιση ε, της αποστολής μας προς τις δύο αυτές ε, χώρες. Ήμασταν εκεί ως ιδιώτες, ε, ως ιδιώτες μας αντιμετώπισαν στην Αλγερία και στην Τινησία, με συγχωρείτε, στην Αλγερία μας δέχτηκαν ως ε, με βυζαντινές ε, ε επισημότητες με πολύ ε, πρωτόκολλο και με λίγα χαμόγελα, ενώ στην Τινησία τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Όμως η Αλγερία ε, σε επίπεδο δημόσιας ε, στάσης είναι πολύ πιο ικανή, ενώ η Τινησία ε, δεν αισθάνεται την ίδια αυτοπεποίθηση. Οι αλγερινή πολιτικοί ε, αισθάνονται, την, έχουν την αυτοπεποίθηση να πούν πως δεν συμφωνούν, ε, πως και οι ίδιοι έχουν πρόβλημα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα εμείς στη Λιβύη, πως πιστεύουν πως την κρίση στη Λιβύη την προκάλεσε η Ευρώπη ε, και οι ομόλογοι μας στην Αλγερία μας τα έξω από τα δόντια. Και όταν του ζητήσαμε κάτι, μα ζήτησαν να του χρηματοδοτήσουμε. Και αυτή ήταν η απάντησή του σε πολλέ περιπτώσει. Οπότε ήθελα να σχολιάσω και αυτή την ε, πτυχή τη ε, επίσκεψη. Κύριε Ζώσνια, σα ευχαριστώ πολύ. Με κάποια θέματα δεν μπορώ πια να συζητώ μαζί σας, Είσαστε ανικανοποιητό. Αλλά για την Αλγερία να σα πω πώ είχατε την ευκαιρία να πάρετε το λόγο σε κάθε μία από τι συναντήσει. Οπότε ζητούσα το λόγο σα τον έδινα. Και Θυμάμαι ότι αναφερθήκατε στο θέμα της χριστιανικής κοινότητας Αλγερίας. Τα είπατε αυτά. Αυτό το λέω για να σας διορθώσω. Γιατί δεν νομίζω πως το σχόλιο αυτό ήταν 100% δίκαιο. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξης που είναι το 9. Συμφωνία με τη Μολδαβία. Εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται, μια και θα πρέπει να φύγω. Έχω την πτήση μου. Νωρί σήμερα. Όντω, να σα ε, ομολογήσω ότι δεν περίμενα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση για την εφαρμογή τη συμφωνία Σύνδεσης με την ε, Μολδαβία. Λάβαμε ωστόσο 182 τροπολογίες. Πολλέ. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, η πιο πολλέ και από πολλές ε, εκθέσεις για πιο μεγάλες χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε την έκθεση πρόοδου και ουσιαστικά η βασική γραμμή κατά την κατάρτιση της έκθεσης είναι ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας ε, διακυβεύεται σοβαρά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχεδόν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο λαό τη ε, Μολδαβία. Μάλλον οι Μολδαβοί δεν πιστεύουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό λοιπόν αυτό μόνο πάτη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα πολιτικά ορόσημα, όχι από γενικέ γενικόλογε υποσχέσει. Γι' αυτό λοιπόν λυπούμαστε για τι πρόσφατε αποφάσει των Μολδαβικών αρχών σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά πρότυπα, αλλαγέ στον κώδικα σε ό,τι αφορά και τις συστάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ε, μας ανησυχεί το θέμα της έλλειψης ανεξαρτησίας του δικαστικού στόματος και η πολύ περιορισμένη πρόοδος που έχει σημειωθεί για τη δίωξη των υπευθύνων για μια απάτη ύψους ενός ε, δισεκατομμυρίου δολαρίων ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ε, μέσων ενημέρωση. είναι μονοπωλιακή δυστυχώ η κατάσταση, είναι στα χέρια κάποιων ορισμένων λίγων. Και συνάδουν, τα όσα αναφέρουμε, με τα ψηφίσματα μας τα προηγούμενα του Ιουλίου του τρέχοντος έτους ε, για την πολιτική κρίση στη Μολδαβία, μετά τις εκλογές στο Κίσνιο, της 4 η Ιουλίου του 2017 για την παροχή μικροχρηματικών πολιτικής ε, ε υποστήριξη προ τη Μολδαβία και στο Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, με χαρά μου διαπίστωσα ότι ήταν πολύ αποτελεσματική η συνεργασία με τις μεγάλες πολιτικές ομάδες. Δεν θα έλεγα βέβαια με όλους και όλες τις ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα μας εξηγήσουν σε διάφορες ε, περιπτώσεις την αντίρρηση τους, Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι αυτό το κείμενο αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση και για έγκριση. Ευχαριστούμε τον κύριο Στρεβίτσιους, λέει ο πρόεδρος και τώρα να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι που επιθυμούν να κάνουν μια παρέμβαση πρέντα, καλνιέται και κρουστία. Ο κύριος Μποστινάρου, Σαφχάουζερ, αυτή και ο κύριος Καστάλντο. Έξι Ομιλητές, σας παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Πρώτος. Α, είναι ο σκιώδη συζητητή μας ο κύριος Κρουστία. Και ο κύριος Κόλμπατσεφ κατέφθασε. We're just trying to sort out who would like... Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κόβατσεφ, Πρέντα, Κανιέτε, Κρουστία, Κανιέτε, Μποστινάρου, Καστάλντο. Μου ξέφυγε κανεί, Κόβατσεφ. Δύο λεπτά έχετε στην διάθεσή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πολύ και τον ε, κύριο Αστραβίτσιου τον Πέτρα για τι προσπάθειε που έκανε και για την επικοδομητική του προσέγγιση κατά την κατάρτιση των συμβαστικών τροπολογιών που συζητήθηκαν χθε στη συνεδρίαση των σκιωδών. Οι πιο σημαντικέ τροπολογίε από πλευρά τη ομάδα μα ε, ελήφθησαν υπόψη στους συμβαστικούς, ε, στις αλλά η ομάδα μα διατηρεί την επιφυλακτική τη και επικριτική τη στάση έναντι των μολδαβικών αρχών. Δεν έχει σημειωθεί και κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά του, μα δημιουργεί μεγάλες ε, ανησυχίε σε ό,τι αφορά και το τι θα συμβεί στη χώρα τις επόμενες, ε, τον επόμενο καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η προσέγγιση των σοσιαλιστών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μας ε, αρέσει γιατί ουσιαστικά αποδυναμώνει και κάπως απαλύνει τη διατύπωση της έκθεσης ε, για να είναι πιο αρεστή στις αρχές της Μολδαβίας. Δεν μας αρέσουν και δεν υποστηρίζουμε τέτοιες ιστραπολογίες εμείς. Δεν θέλουμε να απαλύνουμε τον επικριτικό τόνο της έκθεσης για μας οι αξίες της δημοκρατίας, του κράτος δικαίου, η ελευθερία έκφραση δεν μπορούν και δεν πρέπει να υπονομεύονται. Και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε διατυπώσεις και τροπολογίες που ουσιαστικά ως στόχο έχουν να αποδυναμώσουν τις επικρίσεις από πλευράς της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου. Τι να πω. Καλή επιτυχία εύχομαι στον εισηγητή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όλων των συναδέλφων και όλων των υπαλλήλων. Ευχαριστώ και Κρουστία από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πιστεύω ότι ο εισηγητή παρουσίασε ένα πολύ καλό κείμενο. Είναι πολύ καλή αυτή η βάση για να περάσουμε το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ομάδα μας παρουσίασε και υπέβαλε κάποιες τροπολογίες. Κοιτώντα λοιπόν ε, τι λένε πολλοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι υπάρχει ο κίνδυνος Αντί αυτή η έκθεση να είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικεντρώνεται στα θέματα συμφωνία σύνδεση, ουσιαστικά θα γίνει ένα είδο προεξαγγελία εν των εκλογών. Όλοι ξέρουμε τι γίνονται στην Μολδαβία, ξέρουμε ότι τα πράγματα απέχουν παρασάγκα από τον τέλεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν, όπω γίνεται και για, σε άλλε εκθέσει ε, για διάφορε χώρε, καλό θα ήταν να αναβληθεί η ψηφοφορία για να μην επηρεαστεί η προεκλογική διαδικασία και οι εκλογέ οι ίδιε. Αυτό είναι προ το συμφέρον τη Μολδαβία και είναι και προ το συμφέρον α, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το κύρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη Μολδαβία. Ελπίζω να μην υποστηρίξουν οι συνάδελφοι, γιατί τα συμφέροντα τη Μολδαβία και των πολιτών τη Μολδαβία είναι να παραμείνουν σε μια ευρωπαϊκή τροχιά. Αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί και αυτό θα πρέπει να αποτελεί και το γνώμονά μα ε, σε όλες μας τις πολιτικές δράσεις. το Κοινοβούλιο λοιπόν είναι δυνατό όταν μιλάμε μία φωνή. Το ξέρουμε αυτό. Επανειλημμένα έχει φανεί. Να έχουμε υπόψη ότι δεν θέλουμε να αντικαταπτρίζονται οι εντάσεις και τριβές στη Μολδαβία, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο κύριο Καστάλντο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για τις τροπολογίες. E να σας πω πως είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση εκεί και είναι πολλά τα στοιχεία που συγχωνιγόρουν προς αυτό για το κράτος δικαίου, για την ανεξαρτησία των μίντια και ήμουν εκλογικός παρατηρητής πριν από κάποια χρόνια στις προεδρικές εκλογές στη χώρα και στην συνέντευξη τύπου για πρώτη φορά δεν μας έκανε κανείς καμία ερώτηση μετά τη δική μας ανακοίνωση και το θεωρώ σημαντικό. Λυπάμαι που σε ε, προσωπικό επίπεδο δεν ήμουν παρόν στους σκιώδεις χτες Ίσως ήταν πολύ έντονη αυτή η συζήτηση εκεί και θα ήθελα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την επικοδομητική κριτική. Λάβετε όμως υπόψη και το χρονοδιάγραμμα γιατί θα γίνουν εκλογές στη χώρα και νομίζω πως θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι καλό εμείς να αναβάλουμε την ψήφιση της έκθεσης για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση για το θέμα της Μολδαβίας και δεν νομίζω ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας είναι καλό να χρησιμοποιηθεί ως ε, όπλο στην ε, προεκλογική εκστρατεία αν εμείς λίγο πριν τις εκλογές έχουμε ψηφίσει αυτή την έκθεση. Έχουμε κοινό δρόμο να διανύσουμε με πολύ σημαντικά μηνύματα και θα πρέπει ό,τι κάνουμε να είναι επικοδομητικό και να μην δημιουργήσει περισσότερη πόλωση στα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να τους δώσουμε τα κίνητρα για να κάνουν τη δουλειά τους. Και θα συνεχίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την συγγραφή της έκθεσης. Ε, Ο κύριος Πρέντα. Euh, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας και να σας πω πως εμείς θα τον στηρίξουμε σε όλους τους συμβιβασμούς. Έχω κάποιες από τις τροπολογίες που κατέθεσα και θα ήθελα να τις εξηγήσω και να σας πω για μια φορά ακόμα ποια είναι η κατάσταση στη χώρα. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή πως η κυβέρνηση, η Βουλή, ο τύπος και η δικαιοσύνη κατευθύνονται όλοι από έναν ολιγάρχη ο οποίος δεν έχει στηρίξει από το εξωτερικό, μόνος που τον στηρίζει είναι οι σοσιαλοδημοκράτες των ε, Ρουμάνων δεν έχει άλλη στήριξη από την Ευρώπη και αυτή τη φαντασίωση την πουλάει στην ε, Μολδαβία, γιατί όπως σα είπα δεν υπάρχει ανεξαρτησία του τύπου, είναι όλη από την κυριαρχία αυτού του ανθρώπου. Εμείς εγκρίναμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση, δεν θα χρηματοδοτήσουμε ως Ευρώπη όσο οι δημοκρατικές συνθήκες δεν έχουν ε, επανα ιδρυθεί είναι ένα ολιγαρχικό καθεστώτος μη διάφανο από ολιγάρχες που στηρίζονται από τη Ρουμανία που είναι κράτος μέλος με φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται. Και είμαστε, μπορώ να μιλήσω για μια τρέλα με επιθέσεις οι οποίες προωθούνται στο κοινό και τα οποία όλα αυτά συμβαίνονται στο Κισινιόφ είτε στη Βούκ στο Βουκουρέστι. Μιλάμε για την απόλυτη φαντασία. Αν δεν έχουμε πραγματικές δημοκρατικές συνθήκες στη χώρα, δεν θα πρέπει να στηρίξει η Ευρώπη. Και το γεγονός ότι αναβλήθηκαν οι εκλογές, γιατί το, το θέλει ο κύριος Πλαβότνικ, είναι ένα μήνυμα ξεκάθαρο το τι γίνεται στην πρωτεύουσα σε σχέση με την Ευρώπη. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που το βλέπω. Ευχαριστούμε τον Κρίστιαν Πρέντα και τώρα περνάμε στον κύριο Μποστινάρου. Για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω την πρόταση που έκανε ο εισηγητή μας να αναβληθεί η ψηφοφορία και έτσι να επιτρέψουμε στους κοιόδε εισηγητέ να συνάψουν μια συμφωνία η οποία θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τις δικές μας ε, σύμβολες, γιατί με τέσσερις εξαιρέσεις δεν υπάρχει ούτε μία τροπολογία σοσιαλιστών και δημοκρατών που να έχει μπει στις συμβαστικές. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Ύστερα, τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η Μολδαβία αποτελεί άλλο ένα πεδίο μάχης ε, του ΕΛΚΑ ή θέλουμε επικοδομητικά να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού στην φάση πριν από τις εκλογές. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον επιθυμούμε να δώσουμε το δελτριώδες μήλο προς τους φίλους του ΕΛΚΑ στη Μολδαβία. Μπορούμε πλειοψηφικά, αλλά μην ξεχνάτε ότι το κάναμε και στην περίπτωση του Περίσα και το κάναμε επίση και στην περίπτωση του Και ξέρετε πολύ καλά πώ κατέληξε αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, Πρόεδρε, Σα καλώ ένθερμα να λάβετε υπόψη το ενδεχόμενο αναβολή τη ψηφοφορία προκειμένου να επιτρέψουμε να διεξαχθούν νέε διαπραγματεύσει για να πετύχουμε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό για την έκθεση αυτή. Είναι υπερβολικά απλό, απλοϊκό να ακολουθήσουμε αυτή την οδό και μετά να δρέψουμε τους καρπούς της ε, διχόνοιας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποστινάρου. Δύο λεπτά η Ρεμπέκα Χαρμεσά. Και βέβαια μπορεί κανείς να ζητήσει πάντοτε αναβολή ψηφοφορία και νέες διαπραγματεύσεις. Όμως κάτι που δεν θα ήταν σωστό σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συνδεδεμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, χώρες εταίρους εν τέλει, και βέβαια υπάρχει εγκύτητα προς τις κυβερνήσεις κομματικών σχηματισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή η εγκύτητα δεν θα πρέπει να θολώνει την εικόνα. και ειδικώ στις συζητήσεις και στις ε, χώρες εταίρους, αλλά και εδώ. Ειδικά τώρα για την δημοκρατία της Μορδαβίας οφείλω να πω ότι οι αρνητικές αυτές τάσεις δεν είναι τίποτε το νέο. Από τότε που έγινε η μεγάλη απάτη, απάτη ε, ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, έχουμε στη Μολδαβία πια μια εξέλιξη αρνητική. Ε, είδαμε αλλαγή φρουράς στο Κοινοβούλιο που πραγματικά εκπλήσει. Είδαμε και τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, όπως τη μία αναγνώριση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην ε, πρωτεύουσα Κισινάου, είδαμε βίες διαδηλώσεις, η βίαιη καταστολή διαδηλώσεων, είδαμε να οργανώνονται νέες εκλογές υπό νέο εκλογικό νόμο, όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ε, κριτική και μάλιστα δικαιολογημένη. Νομίζω ότι δεν βγαίνουμε ε, με καθαρή εικόνα από αυτές τις ε, συγκρούσεις εάν προσπαθούμε να επηρεάσουμε συμμαχίες με κυβερνητικά κόμματα. Η έκθεση, έστω να γίνει αναβολή της ψηφοφορίας, η έκθεση όμως πρέπει να είναι ειλικρινής και έντιμη δεν μπορεί να αγνοεί τις εξελίξεις αυτές που έχουν ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτήρα μόνο και μόνο διότι έχουμε εγκύτητα προς κάποιου σχηματισμούς στην κυβέρνηση. Ε, ευχαριστώ. Τώρα, Καρνιέτε Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καρνιέτε. Κυρία Καρνιέτε, θα μιλήσω όμως λετωνικά, κύριε Πρόεδρε, προσοχή, φορέστε ακουστικά. Ε, ε, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες του κύριου Αστοβίτσιους για τη σύνταξη της εκθέσεως που να απηχεί τη γονατική κατάσταση στη Μολδαβία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάθε λόγο να ανησυχεί ε, σχετικά με την πορεία της Μολδαβίας προς την Ευρώπη. Με την έκθεση θα πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Κατ' ουδένα τρόπο επιτρέπεται το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την αναβολή της προφορίας της εκθέσεως, διότι αυτό θα σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές ακολουθούν τις ε, επιθυμίες του ολιγάρχη, του οποίου η νίκη στο Κίσινεβ και την ανατροπή των εκλογικών αποτελεσμάτων δείχνουν ότι δεν υπάρχει ούτε ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, μόνο η άποψη του ολιγάρχη. Και αυτή η απάτη του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ουδής κατέληξε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ούτε έχει το δικαίωμα να τοποθετείται η δημοκρατική αντιπολίτευση. Η μακροοικονομική υποστήριξη προς τη Μοδαβία και οι πληρωμές που γίνονται θα μπορέσουν να, ε, συνεχί... να αρχίσουν και πάλι μόνο όταν θα γίνουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές και υπό τον όρο ότι θα είναι ε, θα είναι νόμιμες εκλογέ αυτές σύμφωνα με τις αρχές του διεθνού δικαίου. Ευχαριστώ κυρία Καρνιέτε. Κυρία Γκόμε, δύο λεπτά παρακαλώ το πολύ. Ε, κυρία Γκόμες, έχω λάβει επισκέψεις από διαφόρους Μολδαβούς που μου έδωσαν μια εικόνα της καταστάσεως εκεί που πραγματικά ε, δείχνει ανατροπή του κράτους δικαίου και βαριές παραβιάσεις μίλησα με εκλεγμένο δήμαρχο ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να καταλάβει την θέση του. Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό σε μια χώρα όπου θέλει εν πάση περιπτώσει να είναι συνδεδεμένη χώρα με την Ευρώπη. Έχω μιλήσει με ανθρώπους για τις ε, διακλαδώσεις αυτής της απάτης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό πραγματικά ότι δεν έχει λάβει χώρα καμιά διαρεύνηση, δεν έχει κληθεί κανεί ενώπιον τη δικαιοσύνη. Είναι καθήκον μα εν τέλει να ασκήσουμε πίεση. Και αυτό θα πρέπει να απηχείται και στις αποφάσεις που θα λάβει το Ευρωκοινοβούλιο. πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα δυστυχώς προηγουμένως να σημειώσω τον κύριο Σαφχάουζερ, ο οποίος λαμβάνει τελευταίο τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για μια φορά και εγώ θα συμφωνήσω με την έκθεση του κύριου Αουστρεβίτσιους και με τον κύριο Πρέντα. Αν και θεωρούνται από τον κύριο Σόρος άνθρωποι ασφαλείς και σίγουροι, που εγώ δεν είμαι, για αυτόν, για τον Σόρος, θα πρέπει να γίνει διαρεύνηση της υπόθεσης του δισεκατομμυρίου και ιδίω όλων των ροών ανακύκλωσης. Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα και με εκπλήσουν που δεν τα, που δεν τα βλέπω και στα ε, και για το πώς ανακυκλώθηκε αυτό το δισεκατομμύριο. Και το μόνο που ζητώ από τους συναδέλφους είναι να μην χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάνε καλύτερα τα πράγματα στο Κόσοβο ή στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά ε, το που εξαφανίζονται τα χρήματα, αλλά και για η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι θα κάνει η πολιτική μου ομάδα. Εγώ πάντω θα υποστηρίξω την έκθεση. Σα ευχαριστώ. Okay. Thank you. σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ενθουσιώδη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Κύριε Αστρεβίτσου, θέλετε πραγματικά την τελευταία τελευταία λέξη. Επιτρέψτε μου να κάνω εγώ πρώτα κάποιες παρατηρήσεις. Ναι. Παρακολούθησα προσεκτικά τα επιχειρηματά σας πολλά στρέφονται γύρω από το ερώτημα αν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Αυτό θα το κρίνουν οι πολιτικές ομάδες. Ωστόσο, εγώ να σας ενημερώσω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει συμφωνηθεί προεξαμήνου. Και το χρονοδιάγραμμα αυτό λαμβάνει υπόψη και το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια μετά τις εκλογές στη Μολδαβία. Δεν είναι δυνατόν. Το άλλο επιχείρημα είναι ότι το χρονοδιάγραμμα που ομόφωνα ψηφίσαμε συντονίζεται με, το, με τις εργασίες στην ε, Γεωργία και Ουκρανία. Άλλο ένα επιχείρημα αυτό. Σας υπενθύμησα εγώ ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Εμπιστεύω με τον κύριο Αστραβίτσιους και θεωρώ ότι θα μπορέσει να βρει μια λύση που να μπορέσει να ικανοποιήσει και τις ανησυχίες όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Ορίστε, για να βρει κανεί λύση στην ε, Μολδαβία θα πρέπει ίσω να κατέβει υποψήφιο στη Μολδαβία. Θα προσπαθήσω να βρω μια λύση. Πάντω, κύριε Ρόεδρε και κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική συζήτηση και τα στέρεα επιχειρήματα που προβάλλατε. Έχουμε μπροστά μα εκλογέ στη Γεωργία. Όμω, ωστόσο, ωστόσο, μάλλον, μέχρι τώρα δεν άκουσα τίποτα για την ε, έκθεση στην Γεωργία. Θυμηθείτε εκείνο το ε, σύνθημα του Κλίντον, η οικονομία ανόητε. Όχι, οι αποφάσεις είναι λάθος στην περίπτωση αυτή. Η κατάσταση στη Μολδαβία η ίδια είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε η προσφορά που θα κάνω ως λύση είναι να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια πιο ενοποιημένη στάση. Θα οργανώσω άλλη μια συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω να είναι παρόντι, παρόντες οι ίδιοι ευρωβουλευτές και όχι οι σύμβουλοι τους, ας αναλάβουν την πολιτική τους ευθύνη. Λοιπόν, πολύ. Εγώ πραγματικά ευνηδιάστηκα όταν κάποιες πολιτικές ομάδες εκπροσωπήθηκαν από συμβούλους. Ανθρώπους, ικανού μεν, αλλά δεν είναι οι υπεύθυνοι βουλευτές αντικρίσουμε λοιπόν κατάματα την πραγματικότητα, όχι αναβολή ψηφοφορία, αλλά άλλη μια συνάντηση των σκιωθών. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο, άλλη μια συνάντηση των σκιωθών. Σα παρακαλώ λοιπόν, ρυθμίστε τα. Για την ώρα προβλέπεται ε, η ψήφιση στις 9 Οκτωβρίου. Κρίστιαν Πρέντα. Α, όχι, ο κύριος Μποστινάρ. Με συγχωρείτε, έχω ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε έχετε την ευγενική καλοσύνη ε, να καθησυχάσετε κάποιους συναδέλφους μας που τους κατέχει μια μανία. Εν πάση περιπτώσει, ανακαλέστε τους την πειθαρχία. Εδώ πραγματικά είναι ντροπή. Ναι, ήθελα να φτάσω στο υπαρθμό 10, λέει ο πρόεδρος, την ε, Γεωργία. Είδα όμως ότι μόλις συζητείτε εδώ η Μολδαβία, ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Επιτροπή Εξωτερικών. Τώρα ίσως να μπορέσουμε να ρίξουμε πάλι τη θερμοκρασία, διότι ερχόμαστε στο υπαρθμό 10, και χωρίς παραπέρα λόγια δίνω τον λόγο στον κύριο Μάμικινς. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ενημέρωση σύντομη για το πώς εφαρμόζεται η Συμφωνία Σύνδεσης με την Γεωργία. Ξέρετε και εσείς πως είναι η πρώτη σχετική έκθεση και πιστεύω πως είναι ακόμα πιο σημαντικό να είναι μία έκθεση με πρακτικά στοιχεία και συγκεκριμένες συστάσεις έτσι ώστε η κοινή μας προσπάθεια να είναι πιο αποτελεσματική. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι γιατί συνεισφέρατε με τις δικές σας τροπολογίες στην έκθεση και αυτή τη στιγμή είναι 229 τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι και επίκαιρο το θέμα αυτή τη στιγμή Κοιτάω τους ε, συμβιβασμούς που θα πούμε, θα συζητήσουμε στις 3 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο με τους Σκιώδης και είμαι σίγουρος πως θα καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό να βρούμε τη συνένεση. Έχουμε πολλές τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την καλή διακυβέρνηση, με τη μάχη κατά της ε, διαφθοράς, τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και με χαρά βλέπω πως τα περισσότερα σχόλια υπογραμμίζουν την ε, πρόοδο που έχει επιτύχει η Γεωργία από τη στιγμή που ετέθησε εφαρμογή συμφωνία. Περιμένω την ε, αποδοτική συνεργασία μαζί σας για να κλείσει η έκθεση και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Μαμίκενς. Πάντα είστε σύντομος. Σκιώδης. Ms. Harms, Castaldo, Gala, and Ms. Kalniete. Okay? We start with Christian. Λοιπόν, ο Κριστιαν Πρέντα, ευχαριστώ πολύ να πω πως ε, στέτινα, ο στέτινα είναι ο σκιώδης, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να μεταφέρω πως είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν έχει ακόμα συμβαστικές προτάσεις, άρα δεν έχουμε μεγάλη πρόοδο. Προσωπικά να σας πω πως κατέθεσα τροπολογίες, οι οποίες υπογραμμίζουν κάποια θέματα και την γενικότερη ιδέα της ενίσχυσης συνεργασίας με τη Γεωργία. Επίσης υπογράμμισα τη σημασία να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το τόσο φιλόδοξο θεματολόγιο που θέλει να απολυτικοποιήσει τους κυβερνητικούς θεσμούς, τους κρατικούς θεσμούς, έτσι ώστε η μη διάφανη διακυβέρνηση και η, ε, η επιρροή η εξοκυβερνητική στις αποφάσεις να εξαλειφθούν έχουμε κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που είναι πολύ σημαντικές και έχουν να κάνουν, και έχουν να κάνουν με την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία συμφωνούν και οι γεωργιανοί ε, φίλοι. Τροπολογίες μου για τον τύπο ε, έχουν να κάνουν με την ανάγκη να υπάρχουν ανεξάρτητα μίντια, να μην εκφοβίζονται οι δημοσιογράφοι και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στη χώρα αυτή όπως και σε άλλες περιοχές με ελευθερία γιατί καμιά φορά λαμβάνουμε μηνύματα δεν θα έλεγα εκφοβισμού ή απειλών αλλά πιέσεων από τα πολιτικά κόμματα. Thank ευχαριστώ πολύ. Είμαι τυχερή γιατί παρακολουθώ το θέμα της Γεωργίας από τότε που είχα πάει το 2016 ε, για την, ε, ως παρατηρήτρια στις εκλογές και είμαι και στη σχετική ομάδα εργασίας για τα, τις δημοκρατικές εκλογές και βλέπω πως η κατάσταση ναι, εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, υπάρχει μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών, αυτό κάνει τεράστια διαφορά και η εταιρική σχέση μαζί μας είναι πολύ σημαντική για την κοινωνία στη Γεωργία. Πολλά προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαστε υπεύθυνοι να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και να βοηθήσουμε τους γεωργανούς οι οποίοι πραγματικά επιθυμούν να αλλάξουν. Θα έλεγα, και εδώ αγγίζω πολλές από τις ερωτήσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι και που υπάρχουν στην έκθεση, και μετά όσα είπε ο συνάδελφος κύριος Πρέντα, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένας χώρος στον οποίο εμείς μπορούμε να φέρουμε τη διαφορά. Γιατί όσο ζωντανή και να είναι η κοινωνία των πολιτών, όσο πλουραλιστικά και να είναι τα μίντια, έχουμε ας πούμε την, ε, ε, την ε, ε, online εφημερίδα που είναι το Ρουστάβι που αναφέρει ε, πολύ συχνά τις ε, απόψεις της αντιπολίτευσης και του κόσμου στην Γεωργία και στην Τυφλίδα, αλλά δεν φτάνει. Αν όλα αυτά σε επίπεδο δικαιοσύνη δεν λειτουργούν, αν υπάρχει ατιμωρησία Εγώ ήμουν την περασμένη εβδομάδα στη Γεωργία, συναντήθηκα με ΜΚΟ και οργανώσει πολιτών και όλοι μοιράστηκαν μαζί μου αυτό το οποίο μοιράζομαι μαζί σας, το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά μου ανέφεραν και διάφορες περιπτώσεις ατιμορρησίας, για παράδειγμα των υπηρεσιών ασφαλείας, που είναι σοβαρά τα πράγματα και δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση ενός νέου που δολοφονήθηκε σε μια επιχείρηση αντιτρομοκρατική εκεί που ζουν ε, οι Τσετσένοι. Και αυτό δημιούργησε προβλήματα γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους. Επίσης, διαφθορά. Πολύ σημαντικό. Και εκεί θα πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Και επίσης είδα πως ε, έχουμε τα κρυπτονομίσματα που δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχει το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα, αλλά είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη διαφθορά να εξαπλώνεται. Θα κλείσω λέγοντας πως οι εκλογές, οι προεδρικές, οι οποίες ακολουθούν, θα είναι ενδιαφέρουσες, ενδιαφέροντες υποψήφοι. Κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο και είμαι τυχερή. Συνάντησα δύο από του υποψηφίου τη αντιπολίτευση και μου είπαν πω κατάφεραν να κάνουν εκστρατεία σε όλη τη χώρα και τα λοιπά χωρί προβλήματα, οπότε αυτό έπρεπε να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Η κυρία Χάρμ έχει το λόγο. Και μην υπερβείτε το χρόνο σας. Ε, ναι, θα συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα με την κυρία Αναγκόμες. Υπάρχουν θετικέ εξελίξεις στη Γεωργία. Και θα ήθελα να μιλήσουμε όχι μόνο για την προετοιμασία των εκλογών, αλλά και για τις ε, πρόσφατες διαμαρτυρίες πριν το καλοκαίρι, ότι η αντιμετώπιση αυθονών ήταν πολύ διαφορετική από ότι στη Μολδαβία και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του καθεστώτος μετά από πίεση του κοινού, η κυβέρνηση θεωρώ ότι τηρεί πιο υπεύθυνη και λογική στάση. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τον τύπο, σε ό,τι αφορά την όλη συζήτηση για το Ρουστάβι 2. Αυτό κατέδειξε ότι είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Γεωργίας και με την αντιπροσωπεία τους εδώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν κοφεύουν στη Γεωργία. Υπάρχει μια κάποια κίνηση και μετακίνηση. Σε ό,τι αφορά και τις μυστικές υπηρεσίες και τη μεταρρύθμιση αυτών, είναι σημαντικό αυτό που ανέφερε η Άννα Γκόμες. Και αυτό έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται, θεωρώ, στην επιρροή της Τουρκίας. Έχω λοιπόν καταθέσει σχετικές τροπολογίες για το θέμα και των διεθνών ε, σχολείων στη Γεωργία, στη Μολδαβία και στην ε, Ουκρανία. Είναι σημαντικό λοιπόν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και το Κοινοβούλιο γενικότερα να παρακολουθούν το θέμα αυτό τακτικά σε ό,τι αφορά την επιρροή της Τουρκίας, η οποία οδηγεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τέσσερις αυτές χώρες και απαγωγέ και στη Μονταβία και στην Ουκρανία και στη Γεωργία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο σε ό,τι αφορά την επιρροή και την πίεση που από την Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μίχελ Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε η συνάδελφο ε, Γκόμε και η συνάδελφο Χάραμ. Για το τελευταίο αυτό θέμα που αναφέρατε, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έω τώρα αντιστάθηκε στην πίεση της ε, Τουρκίας σε ό,τι αφορά την έκδοση του Πρόεδρου. Αφετέρου, συν, συγκρίνοντας την κατάστασή της Γεωργίας με τη Μολδαβία, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει σύγκριση, γιατί είναι σαφώς, σαφές ότι είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο η Γεωργία. Παρά το γεγονός ότι και εκεί υπάρχει ένα άτομο, ένα πολιτικό με σημαντικό πόστο στο πολιτικό κόμμα, χωρί να είναι εκλεγμένο όμω. Δεν συγκρίνεται όμω η κατάσταση. Στη Γεωργία, όπω και στην Ουκρανία, τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα από ποσοτική άποψη σε σχέση με το παρελθόν. Να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά πραγματικά ζούμε καιρού πολιτική ε, πόλωση. Ε, και εγώ από πλευρά μου συχνά έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Βλέπω λοιπόν ότι εισακούεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το σημειώνω ως θετική παρατήρηση. Και ίσως εν ώψη και της ε, πόλωσης της πολιτικής αυτής που υπάρχει και στην αξιολόγηση της κατάστασης του τύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητες πηγές ως σημείο αναφοράς τους δημοσιογράφους ε, χωρίς σύνορα ενδεχομένω ή τις αξιολογήσεις Freedom House ε, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Γιατί εκεί τουλάχιστον έχουμε κάποια αντικειμενική εγγύηση ως προς τις αξιολογήσεις που γίνονται και ίσως λοιπόν στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί και το κείμενο της έκθεσης και των τροπολογιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Μιχαήλ Γκάλερ και το λόγο έχει τέλος ο κύριος, η κυρία Καλνιέτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω λεπτονικά. Βάλτε αν θέλετε τα ακουστικά σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε σχέση με τη Μολδαβία η Γεωργία είναι σε πολύ καλύτερη θέση και σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ε, γιατί οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν, η δημοκρατία φαίνεται ότι λειτουργεί. Οι βασικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαστικό σώμα και στο νομικό σύστημα καθυστερούν ωστόσο. Και το θέμα των πολιτικών κομμάτων φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση η οποία έχει μεγάλες συνέπειες. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε διεθνείς οργανώσεις Δεν είναι δυνατόν να προσχωρήσει κανεί κάποια χώρα αν δεν υπάρχει σαφή ε, διάκριση των εξουσιών σε κρατικό επίπεδο. Και η πολιτική τη ε, Γεωργία θα πρέπει να έχουν υπόψη του λοιπόν ότι χρειάζεται αυτή η διάκριση εξουσιών και θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση των κυβερνών κομμάτων έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η άποψη της αντιπολίτευσης και θα πρέπει να υπάρχει αντίκτυπος της άποψης της αντιπολίτευσης στα πολιτικά κεκτενόμενα. Θα πρέπει να εκπροσωπούνται και αυτοί οι ψηφοφόροι. φέτε επίσης ε, το θέμα των μέσων ενημέρωση. Είναι απαράδεκτο το τι συμβαίνει και θα ήθελα να πω κλείνοντα ότι η Γεωργία έχει πολλά ακόμα να κάνει για να φτάσει σε ένα πραγματικά δημοκρατικό καθεστώ σε ό,τι αφορά τον τύπο, τα δημοκρατικά κόμματα, σε ό,τι αφορά και του όσου επικρίνουν την κυβέρνηση στον τύπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Μαμίκιν, θέλετε να πάρετε το λόγο να τα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις σας. Θα λάβω υπόψη τις τοποθετήσεις σας σε ό,τι αφορά και την ε, μελλοντική συνεργασία μας. Θα λέμε την άλλη εβδομάδα, 3 Οκτωβρίου. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ε, 9 ε, ναι, Οκτωβρίου θα λάβει χώρα η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μα, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Στην Ολομέλεια το θέμα θα περάσει είτε τον Νοέμβριο είτε τον Δεκέμβριο. Και τώρα να περάσουμε στο 11 τη ημερησία διάταξη παρουσίαση συγκριτική μελέτη. Α, ο κύριο Γκάλερ θέλει το λόγο πρώτο. Ε, ναι, επιτρέψτε μου να πω το εξή. Με ενημέρωσαν ότι ο πρόεδρο της Επιτρο... η πρόεδρος μάλλον της Επιτροπής Ενοποίησης του Γεωργικού Κοινοβουλίου είναι μαζί μας εδώ πίσω. Ίσως θα έπρεπε και επίσημα να τη χαιρετήσουμε και να την καλωσορίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Μάλιστα. Μόλις ε, καταφτάσατε. Καλώ ορίσατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είσαστε τακτική επισκέπτρια τη Επιτροπή μα. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα, στην παρουσίαση λοιπόν τη κριτική μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη ενό θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεση στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δεν ε, παρίσταται κανένα από του αντιπροέδρου μα. Αν συμφωνείτε, ποιο θα αναλάβει την προεδρία τη ε, συνεδρίαση, ε, Ρεμπέκα, κυρία Χάραμ, γιατί έχω ένα κατεπήγον τηλεφώνημα το οποίο πρέπει να κάνω και θα επιστρέψω σε 15 λεπτά. Ρεμπέκα, αν θα ήθελες. Okay, thanks uh, for the trust uh, Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, λέει η κυρία Μπέκα. Χάρομες αναλαμβάνω τα ενία της Προεδρίας με μεγάλη μου χαρά, μεγάλη ευθύνη και χαρά να συντονίσω το πάνελ αυτό, γιατί την παρουσιάσαμε αυτή τη μελέτη ήδη σε ένα διαφορετικό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συζητήσαμε και πρόσφατα στο Κίεβο. Έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω τον καθηγητή, την καθηγητρία Κατερίνα Βολτσούκ από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, η οποία εκειδικεύεται στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, μετασοβιετικών χωρών στα πλαίσια της πολιτικής εταιρικής γειτονικής σχέσης. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι στις 30 Αυγούστου λάβαν χώρα τρεις μελέτες για το επίπεδο προσέγγισης ε, των συμφωνιών σύνδεσης και σήμερα έχουμε αυτή την τελευταία μελέτη, την οποία ζητήσαμε ως τμήμα των εργασιών μας. Επικεντρώνεται στη λειτουργία των θεσμών στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών. Με άλλα λόγια, το πώς και γιατί εφαρμόζονται κάποια τμήματα των συμφωνιών και κάποια άλλα δεν εφαρμόζονται. Προτού δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Βόλτσουκ να αντράξω την ευκαιρία και να πω ότι οι συνάδελφοι που εργάζονται στην ΑΦΕΤ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, α, αυτές τις εμπειρίες που έχουν συλλέξει από τις διαδικασίες εφαρμογής θα πρέπει να συζητηθούν πιο ενδελεχώς, με έναν πιο εντατικό τρόπο, γιατί η διαδικασία υλοποίηση είναι πολύ πιο απαιτητική και περίπλοκη από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Στην αρχή των φιλόδοξων αυτών των προγραμμάτων. Για μένα λοιπόν ήταν αρκετά σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι υπό δύσκολε συνθήκε σε αυτές τις τρεις χώρες υπό επίθεση από τη Ρωσία σε διαφορετικούς βαθμούς, γιατί η Ουκρανία αντέχεται μεγαλύτερες πιέσεις από τι υπόλοιπε χώρες, αλλά ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες αυτές, με μία ουσιαστικά δύναμη οικονομική υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε αυτέ είναι σε διαδικασία αλλαγή και μεταμορφώσεις. Κυρία Βόλτσοκ, έχετε το λόγο και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. I have to apologize to the translator. a Slavic speaker. Να ζητήσω συγγνώμη. Με συγχωρείτε που μιλάω γρήγορα, αλλά έχουμε σλαβικής καταγωγής αγορητής. Να σας πω πως έχουμε πολύ εμπειρογνωμοσύνη εδώ, έχουμε ε, καλό θεματολόγιο και εγώ ουσιαστικά δεν ξέρω αν βοηθάω με την παρουσία μου. Θα ήθελα να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και συγχωρέστε με γιατί ίσως ελπίσατε στην παρουσίασή μου, θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Όχι, εγώ μπορώ να συζητήσω μαζί σας θέματα με λεπτομέρειες, αλλά θέλω να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και να εστιάσουμε στο τι ακριβώς σημαίνει η Συμφωνία Σύνδεσης για τις χώρες αυτές σε επίπεδο εφαρμογή. Και να σας πω πως εδώ κυρίως έχουμε να κάνουμε με το συντονιστείτε ή χαθείτε. Είναι περίπλοκες, εξαιρετικά περίπλοκες συνθήκες, από τις πιο περίπλοκες που υπάρχουν παγκοσμίων και συνάπτονται με χώρες οι οποίες βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα πολιτικού, νομικού ε, και ε, κοινωνικού κύκλου. Άλλα επίπεδα ανάπτυξη, τεράστια πρόκληση και στη μελέτη έκανα μία πολύ προσεκτική απογραφή των όσων συμβαίνουν. Ποιοι θεσμικοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν στην εφαρμογή. Γιατί έτσι μας δίνει η επισκόπηση αυτή μία δυνατότητα να καταλάβουμε αν οι χώρες είναι σε θέση να συμμορφωθούν και να ε, εφαρμόσουν την συμφωνία μέσα στις ε, χρονικές ε, προθεσμίες. Το πεδίο εφαρμογή μελέτης το περιγράφω. Δεν πρόκειται να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, είναι όμως μία επισκόπηση και βασίζεται στην προϋπάρχουσα πραγματογνωμοσύνη μου. Και πρέπει να σου πω πως ταξίδεψα και στις τρεις χώρες και συζήτησα πολλά θέματα. Για τους ε, θεσμικούς μηχανισμούς τι ακριβώς έχουμε κατά νου. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία εδώ. Πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, ε, η συμφωνία στηρίζεται στο υψηλότερο ε, πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο σε λόγια, αλλά εάν σπρώχνουν προς την εφαρμογή. Δεύτερον, συντονιστικός μηχανισμός. Στη Βουλή, στην κυβέρνηση, οι υπηρεσίες συντονίζουν τη δράση τους, γιατί πολύ συχνά έχουμε οριζόντια φύσης θέματα. Και το πιο σημαντικό είναι θεσμικό δυναμικό και πολύ συχνά αυτό δεν το βλέπουμε αρκετά και στην Βουλή αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξέρουν τη δουλειά τους και για ποιο λόγο ε, ε, αναλαμβάνουν δράση είναι στις κατάλληλες θέσεις. What we have Στην προηγούμενη συζήτηση συμφωνίες σύνδεσης είχαμε το εξής δύο συμφωνίες σε μία. Έχουμε τη γενικότερη συμφωνία για πολιτική συνεργασία με τον πολιτικό διάλογο, οπότε έχουμε το πολιτικό σκέλος συμφωνίας που τίνει να είναι γενικόλογο, να έχει χαλαρές λίτρες, ρίτρες οι οποίες δεν συνοδεύονται συνήθως από προθεσμίες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν μιλάμε για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, εκλογική μεταρρύθμιση δεν έχουμε συγκεκριμένους δείκτες και συγκεκριμένες προθεσμίες. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική με τα πιο τεχνικά κομμάτια της συμφωνίας και κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με την κλαδική συνεργασία και τις ζώνες ελεύθερου, ελεύθερων συναλλαγών, όπου σε κάποια σημεία έχουμε τεράστιο όγκο λεπτομεριών και αυτές συνοδεύονται από απαρέγκλητες προθεσμίες. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο διαφορετικά σκέλη. Και όταν μιλάμε για τη συμφωνία σύνδεσης, κυρίως εστιάζουμε στο ένα κομμάτι που σας περιέγραψα, στο άλλο, όχι και στα δύο μαζί. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπάρχει μια έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ των δύο, γιατί στη Μολδαβία, για παράδειγμα, έχουμε άλλες ε, μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό επίπεδο και άλλες στο τεχνικό. Και άλλους ρυθμούς. Άρα λοιπόν το πολιτικό κομμάτι είναι σημαντικό και έχει να κάνει με την πολιτική συνένεση για την προευρωπαϊκή προσέγγιση, όχι σε επίπεδο δηλώσεων, επαναλαμβάνω, αλλά με προώθηση των στρατηγικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Και όχι μόνο σε επίπεδο ελίτ, αλλά με την τοποθέτηση προσωπικότητα. Ε, έτσι ώστε να ηγηθούν των προσπαθειών και πολλές φορές ε, με ε, συγκρουσιακή πολιτική που χρειάζεται. Ξέρετε, ο κόσμος έρχεται, ο κόσμος φεύγει. Γενικά, θα έλεγα πως η πολιτική βούληση είναι πιο αδύναμη από την διοικητική προσπάθεια που γίνεται. Σε διοικητικό επίπεδο έχουν γίνει βασικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε μία από τις χώρες αυτές έχουμε τα συντονιστικά όργανα, έχουμε την ενδυνάμωση ε, στο εσωτερικό των Υπουργείων, των αρμόδιων Υπουργείων και στη Βουλή έχουμε κάποια πραγματονόση που δεν φτάνει αλλά αυξάνεται και μία κατανόηση ενδεχομένως πως χρειάζονται πυρογνώμονες. Οι χώρες λοιπόν αναγνωρίζουν ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και έχουν αναλάβει δράση. Ε, έλεγχη συμμόρφωσης, κοινοβουλευτικές επιτροπές, συντονιστικά όργανα, όλα αυτά υπάρχουν. Όμως έχουμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες και το να λειτουργούν σωστά μέσα στους υφιστάμενους πολιτικούς θεσμούς και διαδικασίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε πως στην Ουκρανία η Βουλή έχει θέματα εσωτερικών διαδικασιών και νομοθετικής δραστηριότητας που πρέπει να λυθούν. Άρα λοιπόν πώς να γίνεται καλός συντονισμός όταν δεν είναι πολύ αποτελεσματική η Βουλή. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνει κανείς μόνο εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών αλλά και χρήση αυτών. Και εδώ πρέπει να δούμε αυτό το κομμάτι της μελέτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η θεσμικοί μηχανισμοί να μην λειτουργούν απομονωμένοι, αλλά να αποτελούν μια παγιωμένη τακτική στο όλο πεδίο διακυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σύνδεσης να χρησιμοποιηθεί ως εχμή δόρατος στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, στην χάραξη πολιτικής αλλά όχι με απομονωμένο τρόπο. Οπότε οι γενικότερες αδυναμίες στη χώρα βεβαίως και επηρεάζουν την εφαρμογή της συμφωνίας, ακόμα και στο τεχνικό σκέλος. Τα συντονιστικά όργανα τα πάνε καλύτερα όταν μιλάμε για ε, τα παραρτήματα της συμφωνίας γιατί έχουν και τις κατάλληλες μονάδες που ασχολούνται. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μια διχοτόμηση σε κάποιο βαθμό των δύο διαφορετικών επιπέδων και αυτό μπορείτε να το δείτε και στα σχέδια εφαρμογής. που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα τεχνικά κομμάτια και δεν έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, αλλά με τις προθεσμίες, με τα συγκεκριμένα σχέδια δράσης που έχουμε στη συμφωνία. Αυτές οι δράσεις είναι αυτές τις οποίες εγώ θα χαρακτήριζα εκπαίδευση, σεμινάρια, μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να δούμε τα παραδοτέα και να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι θεσμικές υπηρεσίες στην εφαρμογή των νομικών τους υποχρεώσεων πόσο σέβονται τις προθεσμίες και κατά πόσο επηρεάζονται από τις προθεσμίες, κάτι το οποίο είναι πολύ προβληματικό για τη Μολδαβία και την Ουκρανία, γιατί πολύ συχνά τονίζουν την νομική εναρμόνιση, που είναι ένα μάλλον θολό κόνσεπτ, που είναι ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με το κεκτημένο, αλλά που αποτελεί πάρα πολύ τεχνικό καθήκον που χρειάζεται πολλή ενέργεια με αποτέλεσμα να μην δίδεται η απαραίτητη προσοχή για να γίνεται επιπτωσιολογική μελέτη. Και αν θέλουμε, για παράδειγμα, να έχουμε επιθεωρητές δημόσιας υγείας ή ε, ασφάλειας τροφίμων, πού θα πρέπει να βρίσκονται, πού θα είναι η έδρα τους, πώς θα πρέπει να εκπαιδευτούν, πόσο να εκποδευτουν ποσο κοστιζει το να στήσει κανείς εργαστήρια. Ακόμα δηλαδή και στα πιο τεχνικά κομμάτια, είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται επί τόπου. Όλες οι χώρες το προσπαθούν, αλλά δεν μπορώ να πω πως οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί πλήρως, όπως θα έπρεπε. Έχω την αίσθηση πως πρέπει να επιταχύνω Έχουμε σύστημα υποβολής αναφορών μεν, αλλά όχι ένα σύστημα πραγματικής παρακολούθησης, γιατί τα, ε, υπηρεσίες συντονισμού απλώς συντονίζουν. Δεν έχουν την πολιτική ισχύ να κάνουν κάτι παραπάνω μέσα στη χώρα. Και αυτό που βλέπω είναι μια... Είναι κάποια στεγανά μεταξύ των εθνικών σχεδίων μεταρρύθμισης και των τομεακών αλλαγών και στρατηγικών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση για τις χώρες που πρέπει να ενισχύσουν το δυναμικό τους, να κάνουν και στο δημόσιο κλάδο κάποιες μεταρρυθμίσεις, κυρίως Μολδαβία, Ουκρανία, και αυτό συμβαίνει. Παρόλες τις αρνητικές εξελίξεις ε, στη Μολδαβία, έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά χρειάζεται χρόνος. Και παράλληλα τρέχει ο χρόνος για τη Συμφωνία Σύνδεσης και για μένα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διτή προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς γίνεται η εφαρμογή. Και όταν κοιτάμε στο Κοινοβούλιο, όντως εγκρίνουν τις βέλτιστες και αυτούν τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά όταν έρχεται στις επιτροπές το θέμα δεν είναι πάντα σαφές τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συνδυάζονται με αυτό που κάνουν άλλες ε, επιτροπές και το τι κάνει η Ουκρανία πιο συγκεκριμένα. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να υπάρχουν εμπειρογνώμονες στις βουλές για να έχουν χάραξη πολιτικής και θέσπιση προτεραιοτήτων. Είναι σημαντικό αυτό. Και θέλουν στήριξη, θέλουν βοήθεια όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως από εσάς. Και για την νομική εναρμόνιση είναι πολύ θολό, πολύ ασαφές και έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μελέτη σχετικά. με χαρά να τα ξαναπούμε με περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειάζεται. Ένα πρώτο τελευταίο για την ευρωπαϊκή στήριξη και να σας πω γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή η είδητη προσέγγιση. Γιατί έχουμε αυτή τη στήριξη και πώς μπορούμε να την κάνουμε για να έχουμε καινούριου θεσμούς και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι πολλά κομμάτια της εφαρμογής ε, της συμφωνίας γίνεται μέσω της κλασικής τεχνικής βοήθειας και επειδή το κοίταξα, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται και από μια αξιολόγηση αναποτελεσματικότητας της τεχνικής βοήθειας επιτόπου που δεν προέρχεται από τη διαφθορά ε, και ε, προσπάθειες παράκαμψης ε, της νομοθεσίας, αλλά από υπερβολικά περίπλοκους κανόνες που έχουν ως στόχο την αποφυγή διαφθοράς. Αυτό το οποίο είδαμε στις συζητήσεις και το είπαν και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες και οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι όσοι βρίσκονται επί τόπου είναι το ότι ο συντονισμός και η διαδικασία εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπαρκής. Δεν έχουν το δυναμικό και δεν στηρίζονται παρκούς. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές συστάσεις στη μελέτη μας, πολλές σελίδες με γενικόλογε συστάσει που καλύπτουν όλες τις χώρες και τους ευρωπαϊκούς θεσμού. και επίσης να σας πω πως θα πρέπει να εγκρίνουμε ένα πιο ρεαλιστικό ε, πλαίσιο, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και στρατηγική και να περιμένουμε να οικοδομηθεί το δυναμικό γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα το προσπαθούν αλλά δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν όλες τις δεσμεύσεις τους. Και έχω και συγκεκριμένες διαφάνειες που είναι Χώρα, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, με συγκεκριμένα θέματα, αλλά λέω να μπω κατευθείαν στο συμπέρασμα. Και όπως είπα προηγουμένως, ότι οι βέλτιστες πρακτικές είναι ήδη ευρύτατα γνωστές και γίνονται σημαντικές προσπάθειες να εφαρμοστούν. Όλες οι χώρες έχουν τους μηχανισμούς που χρειάζονται έχουν κάνει πρόοδο. Όχι επειδή ήρθαν αργότερα οι συμφωνίες τους, αλλά επειδή πραγματικά είχαν ε, πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή τους και το είπα και όταν το συζητήσαμε με τις χώρες μου είπαν το προσπαθούμε. it's not geared to address the political aspect of the association agreement. Δεν μπορούμε να δούμε την νομική διάσταση, ε, εμείς όταν συζητάμε με τις χώρες. Είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά υπάρχει και αυτό. Βεβαίως η διακυβέρνηση επηρεάζεται από όλα τα παραπάνω. Η ποιότητα θα πρέπει να βελτιωθεί πριν προχωρήσουμε σε μια εφαρμογή η οποία θα είναι αποδοτική και αποτελεσματική. Το θέμα του δυναμικού του κράτους αυτή τη στιγμή συζητιέται, αλλά ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι χρειάζεται χρόνος. Χρόνια οι προθεσμίες όμως τρέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τεράστια στήριξη και για την Ουκρανία να σας πω πως ήταν ένα καταπληκτικό πειραματόζωο για την ε, αναθεώρηση του τι γίνεται ε, σε επίπεδο οικοδόμησης δυναμικού. Αλλά η τεχνική βοήθεια νομίζω για μένα έχει ξεπεραστεί τουλάχιστον με την τρέχωσή τους μόρφη και δεν είναι πια τόσο αποτελεσματική. Οπότε είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από όλα αυτά, αλλά έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και μια υπερδραστηριότητα στις χώρες αυτές. Είναι όμως τεράστια πρόκληση, όχι μόνο για τις χώρες εταίρους, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο. Νομίζω ότι εντάσσεται καλά στην, ε, ε, σε εκθέσεις εφαρμογής που συζητούμε και οι συγητές και σκιώδεις, ειδικά πριν από τη συζήτηση, μπορούν να εξετάσουν τις συστάσεις που κάνετε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συμμετοχή μας, δηλαδή με τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ε, Euronest, έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμό και στη Euronest προέτους έχουμε ιδρύσει ομάδα εργασίας για την εφαρμογή των συμφωνιών συνδέσεως που είναι από τα μάλλον η ομάδα αυτή είναι από τις πιο σημαντικές μέσες δραστηριότητες της Euronest θα πρέπει να τονιστεί επίσης νομίζω ότι τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων έχουν ιδρύσει ήδη κοινοβουλευτικές συνελεύσεις και τρεις αυτές χώρες δηλαδή, για να, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, για να συνεχίζεται η ανταλλαγή απόψεων. Συμμετέχουν σε αυτά βεβαίως με όλες τις διαφοροποίησεις και επαφίεται σε εμάς τώρα να προβληματιστούμε και για τη δική μας συντονισμένη απάντηση στις επισημάνσεις της μελέτης σας. Επειδή πάμε τώρα και στην δέκατη ε, επέτειο του χρόνου δηλαδή της ανατολικής γειτονίας, θα είναι καλό να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς να περιληφθούν στα έγγραφά μας και τα σημαντικά διδάγματα που αντλήσαμε τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Σάντρα Καλνιέται τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, ιδίω εσά για την πολύ ε, ικανή επισκόπηση ιδίω για τα θέματα των συμφωνιών συνδέσεως. Εκλέγομαι σε μια χώρα που προ 14 ετών, ίσως και περισσότερα, ε, πέρασε από τη διαδικασία αυτή, ενώ τη Λετωνία. Και βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό ένα από τα συμπεράσματά σας, ότι δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά την προσέγγιση χορήγησης τεχνικής υποστήριξης. Η αδίποτε απόφαση στη διαδικασία εφαρμογής μπορεί να έχει ε, βαρύτερες ή λιγότερο βαριές πολιτικές επιπτώσεις στον κόσμο, τον πληθυσμό δηλαδή. Η δε πολιτική βούληση των κυβερνήσεων, των θεσμών τους, του, των κοινοβουλίων, του, μάλλον του κοινοβουλίου μιας συγκεκριμένης χώρας, έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν και συνδέονται πολύ με το επίπεδο γνώσεως που διαθέτουν των διαδικασιών ένταξης. Θα χαρώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ε, διαβιβάσετε ηλεκτρονικά την μελέτη σας στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Πολύ ευχαρίστω θα διαθέσω χρόνο για να την μελετήσω προσεκτικά. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Η κυρία Χάρμ, Προεδρεύουσα, σα ευχαριστώ πολύ. Έχετε άλλε ερωτήσει ή σχόλια. Όχι για την ώρα. Σα δίνω πάλι το λόγο λοιπόν και σα δίνω και χρόνο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι έχω συνεργαστεί στενά με συναδέλφους σας της Λιθουανίας ιδίως και βασίζομαι πολύ στις κρίσεις συναδέλφων από τις ε, ε, χώρες υπό ένταξη ή τι συνδεδεμένε χώρε καλύτερα. Και ένα από τα θέματα, διότι τα γνωρίζουν τα πράγματα αυτά καλά οι άνθρωποι αυτοί, ένα από τα θέματα είναι γιατί στην Μολδαβία ή στην Ουκρανία έχουμε 4 ή 5 γενιέ έργων τεχνική υποστήριξη, ενώ η Λιθουανία είχε μόνο 5 γενιες εργων τεχνικη υποστηριξης ενω η λιθουανια ειχε μονο ενα υπήρχε προεταξιακή συνεργασία με τη Λιθουανία, αλλά δεν υπήρχαν στην Μολδαβία και Ουκρανία, για παράδειγμα. Γιατί λοιπόν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα και δεν διδασκόμαστε από τα σφάλματά μας. Και ίσως, να, ίσως να μην είναι τόσο ε, δίκαιο, ας πούμε, αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά τόσο πολλά πράγματα. Όταν όμως πρόκειται για την τεχνική υποστήριξη, δεν βασίζεται στην πραγματικότητα σε βέλτιστες πρακτικές, έχω αναθέσει μελέτη για την ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και εκεί περιλαμβάνονται πολλά θετικά πράγματα. Υπάρχουν όμως και πολλά φαντάσματα από τη δεκαετία του 90. Το πρόγραμμα τάσης για την υποστήριξη και ορισμένες υποθέσεις αθεμελίωτες για το πώ λειτουργούν οι χώρε αυτέ, που συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο όγκος διεθνού υποστήριξη με εμπειρογνώμονες που πάνω και έρχονται και ε, παρόλα αυτά πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτά αντιμετωπίστηκαν στην Ουκρανία. Στη Μολδαβία όμω, κατά τη γνώμη μου, ίσω αυτή αποτελεί το παράδειγμα, όπου τα πράγματα δεν αποδίδουν το ίδιο καλά, Όπω σε άλλε περιπτώσει, όπω η Λιθουανία, σε ό,τι αφορά τις ε, συνέπειες, τις επιπτώσεις των προσπαθειών όλων αυτών των εμπειρογνωμόνων που πάνε στη Μολδαβία να αλλάξουν τα πράγματα επί τόπου. Πολύ ευχαρίστω να τα συζητήσουμε αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται ε, άντληση διδαγμάτων και stock taking και ότι αυτό έχει καθυστερήσει. Και τονίζω επίσης και τις απόψεις πολλών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμπειρογνώμονε Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εργάζονται επί τόπου και οι οποίοι δηλώνουν ε, ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι ε, σε ό,τι αφορά την πρόοδο που επέρχεται από τις προσπάθειές τους. Ε, σταματώ εδώ με αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συνεχιζόμενη δέσμευσή σας στο θέμα αυτό και για το τελευταίο σας θέμα, στην τελευταία, ή μάλλον στην τελευταία μας αποστολή στην Ουκρανία. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν ότι επενδύουμε πολλά σε εμπειρογνώμονες και τις επισκέψεις τους, των εμπειρογνωμόνων στις χώρες αυτές και διαμαρτυρόμεθα μετά ότι οι θεσμοί δεν αναπτύσσονται όπως θα θέλαμε. Όμως δεν επενδύουμε επαρκώς σε εμπειρογνώμονες εντός των θεσμών ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Αυτή απαιτείται. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές που μας παρέσχετε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να προεδρεύσω θα επιστρέψω ωστόσο τα ενία της συζητήσεως στον ε, κύριο Μακάλιστερ, ο οποίος έρχεται και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ.